Je vous Λοιπόν, να συνεχίσουμε, αν και δεν έχουμε όλους παρόντες, αλλά πρέπει να αρχίσουμε, γιατί δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε περαιτέρω. Το πρώτο θέμα είναι ο Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ασχοληθούμε κυρίως με τα πιλωτικά προγράμματα και τις ε, προπαρασκευαστικές δράσεις. Πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Σούκοβα που είναι Διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μην υπάρχει παρανόηση, να διευκρινίσω τι πρόκειται να κάνουμε τώρα. Σήμερα η συζήτηση θα εστιάσει στα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Αυτά δηλαδή που εγκρίθηκαν κατά τις προηγούμενες ε, κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Οι συντονιστές ήθελαν να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε μια σφαιρική αντίληψη για το πώς ε, οι ιδέες μας μεταφράζονται στα προγράμματα αυτά, στις πιλωτικές δράσεις δηλαδή και στις προπαρασκευαστικές ενέργειες και πώς υλοποιούνται από πλευράς χρονοδιαγράμματος κλπ. Παραλαμβάνω, η συζήτηση που θα κάνουμε τώρα δεν έχει να κάνει με το σχέδιο γνωμοδότησης της ε, συναδέλφου κυρία Κλούν που έχει να κάνει με το σχέδιο προπολογισμού του 2018. Αυτό θα το συζητήσουμε στις 25 Απριλίου με τη συμμετοχή ιδιαίτερα του κυρίου Μούρεσαν που είναι ο εισηγητής μας για τον προπολογισμό. Μεταξύ λοιπόν των διαφόρων προπαρασκευαστικών και πιλωτικών ενεργειών που αναφέρονται σήμερα, έχουμε ιδιαίτερα την ενίσχυση της ε, επιχειρηματικότητας των νέων μεταναστών, υπεύθυνη Γενική Διεύθυνση, είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, στο το πιλωτικό πρόγραμμα ΑΛΕΚΟ, που είναι η δυνατότητα συνεργασίας για την επιχειρηματικότητα, επίσης Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξη, Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την κινητικότητα των μαθητευομένων και τις ε, δεξιότητες για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι δικό μας θέμα και ασχολείται η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης στο πιλωτικό πρόγραμμα για ένα οικοσύστημα που θα επιτρέψει τη συνεργασία των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις και τις πλατφόρμες στην Δυτική Πομερανία και σε κάποιες ε, ε, περιοχές της Υπέθρου στην Πολωνία. Προπαρασκευαστική δράση τώρα για την ε, ενδοκινοτική κινητικότητα των ανέργων άνω των, 25, των 35 ετών, προπαρασκευαστική δράση, εγγύηση για την παιδική ηλικία, εγγύηση παιδική ηλικία και βοήθεια προς την παιδική ηλικία, έμπλη και προπαρασκευαστική δράση για την αξιολόγηση των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας της ανώτατης εκπαίδευσης. Γενική Διεύθυνση, κάποια Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν. Αυτές είναι οι πιλωτικές δράσεις και προπαρασκευαστικές ενέργειες που είναι σε εξέλιξη. Να δώσω το λόγο για ένα δεκάλεπτο, το λόγο στην κυρία Σούκοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας με χαρά να σας παρουσιάσω σύντομα την έκθεση. Έχουμε και ένα PowerPoint. Την πρώτη ενδιάμεση έκθεση την έχουμε ήδη υποβάλει όπου περιγράφουμε όλα τα 79 πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις που θα εφαρμοστούν το 2017. Η έκθεση αυτή καλύπτει χρηματοδοτήσεις 62 εκατομμυρίων για τις προπαρασκευαστικές δράσεις και 40 για την εφαρμογή πιλωτικών δράσεων. Επίσης σας ε, έχουμε υποβάλει αναλυτική περιγραφή των ε, προγραμμάτων αυτών, του περιεχομένου. Έχουμε και χρονοδιάγραμμα για όλα αυτά. Και θα σας παρουσιάσουμε μια δεύτερη έκθεση που θα είναι τμήμα του σχεδίου προπολογισμού για το 18 τον Ιούνιο, τρέχοντος. Τώρα, μόλις είπατε, εντός των αρμοδιοτήτων μας έχουμε ένα πιλωτικό και μία προπαρασκευαστική και μία συμπροματική δράση που είναι η εγγύηση για την παιδική ηλικία. Σας εξηγήσω γιατί δεν ε, ανήκει σε αυτές δύο κατηγορίες λόγω του τρόπου εφαρμογής που προτείνουμε για το 2017. Να σας εξηγήσω το πρώτο πρόγραμμα το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κινητικότητα των μαθητευομένων, ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ε, και ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων. Είμαστε στη δεύτερη χρονιά εφαρμογής. Συνολικός στόχος είναι να διευκολύνει την μακροπρόθεσμη κινητικότητα των μαθητευομένων, εξετάζοντας διάφορες ε, δυνατότητες για να υπάρξει αναγκαία υποδομή κινητικότητας και διάφορες υπηρεσίες, για παράδειγμα στέγαση, μαθήματα εκμάθησης γλώσσας, πρακτικές πληροφορίες και ασφάλιση. Και θα εξετάσουμε τρόπους ούτω ώστε αυτές οι θέσεις μαθητείας να γίνουν πιο ελκυστικές για τους νέους. Αυτό είναι ένας ευρύτερος στόχος της δουλειάς μας. Για να υπάρξει περισσότερο ενδιαφέρον μεταξύ των νέων για αυτές τις ε, θέσεις μαθητείας. Για να μπορέσουν έτσι να ενταχθούν ευκολότερα στην αγορά εργασίας. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, το 2017, θα κάνουμε μια προκήρυξη για τη χρηματοδότηση ενός περιορισμένου αριθμού διευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπου θα συμμετάσχουν βασικοί φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση και τη μαθητεία, αλλά θέλουμε να υπάρξουν και διαμεθοριακές ε, κινητικότητες για να προετοιμάσουμε την πιο μακροπρόθεσμη εφαρμογή ε, μιας ε, υψηλής ποιότητας κινητικότητα, ελάχιστης διάρκειας έξι Έχουμε επίσης και ένα σχέδιο ενημέρωση για τα θέματα αυτά, ούτω ώστε να προσεγγίσουμε και τις εταιρείε και άλλους θεσμούς που θα μπορούσαν να δεχθούν μαθητευόμενους. Φέτος λοιπόν, στις 25 Ιανουαρίου συγκεκριμένα, κάναμε την προκήρυξη για προτάσεις. Προθεσμία ήταν η 29η Μαρτίου για την υποβολή προτάσεων. Τώρα αξιολογούμε τις προτάσεις ούτως ώστε το τρίτο τρίμηνο του 2017 να αρχίσουν να εφαρμόζονται τα προγράμματα. Συνολική χρηματοδότηση 2 εκατομμύριων έχει αυτή η προκήρυξη. Και κάποιες πιστώσεις από το 2016 που μας έμειναν από την προηγούμενη προκήρυξη. 840.000 συγκεκριμένα. Επίσης είχαμε και μία συνεδρίαση ενημέρωση στις 22 Φεβρουαρίου με τους ενδιαφερόμενους φορείς Νομίζω ότι οι προτάσεις που μας έχουν υποβληθεί είναι καλής ποιότητας και θα μπορέσουμε να δεσμεύσουμε και να ταμιεύσουμε όλα αυτά τα ποσά. Επίσης θέλουμε να υπάρξει περισσότερη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητευομένων και αυτό το κάνουμε μέσω μια σειράς υπαρχουσών πρωτοβουλειών, μέσω και της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Μαθητεία, τη στήριξη της Κομισιόν μέσω του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για, Συμφώνου για τους Νέους και επίσης μέσω της εβδομάδας για την επαγγελματική κατάρτιση και τις δεξιότητες που είχαμε το Δεκέμβριο του 2016. Θα γίνεται τακτικά κάθε χρόνο προς το τέλος του χρόνου και κυρίως εστιάζουμε στην ποιότητα της ε, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τώρα μια άλλη πιλωτική δράση που έχουμε στο πρόγραμμά μας είναι επανενεργοποιήσουμε το πρόγραμμα κινητικότητας για ανέργους άνω των 35. Είναι στη δεύτερη χρονιά εφαρμογής και αυτή η δράση. Στόχος να βοηθήσουμε τους μακροπρόθεσμα ανέργους ε, ενήλικε να βρουν εργασία ή θέσει θέσεις μαθητείας σε άλλα κράτη-μέλη. Έχουμε παρόμοια μέτρα όπως και στο παρελθόν και θα επεκτείνουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα περαιτέρω. Το 2016 είχαμε το πρώτο κύμα ε, προτάσεων και προγραμμάτων και η πείρα που έχουμε εξαγάγει θεωρούμε ότι θα μας βοηθήσει σε αυτή τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής. Υπάρξουν και μέτρα στήριξης. Θα επικύλουν ανάλογα με τις αγορές εργασίας. θα δώσουν δυνατότητες σε άτομα να πάνε σε άλλες χώρες, να μάθουν περισσότερες γλώσσες, να τους βοηθήσουν δηλαδή να ενταχθούν και περισσότερο και στη χώρα όπου θα υπάρχει αυτή η μαθητεία. Οι δικαιούχοι θα είναι άτομα, είναι ε, άτομα που προσπαθούν να βρουν δουλειά και που προσπαθούν να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή η δράση Θέλουμε να εφαρμοστεί με απλουστευμένες διαδικασίες γιατί αυτό θα βοηθήσει. Οι θέσεις μαθητείας που θα παράσχουμε θα πρέπει να έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών μηνών και μέγιστη έξι μηνών. Η απόφαση για την εφαρμογή του 2017 για την χρηματοδότηση ενεκρίθη στις 22 Μαρτίου και προετοιμάζουμε την προκήρυξη για προτάσεις που θα δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες. Στόχος μας λοιπόν είναι τα προγράμματα να ξεκινήσουν το τελευταίο τρίμηνο του 2017 ή το αργότερο το πρώτο τρίμηνο του 2018. Θέλουμε να υπάρχουν όμιλοι από τουλάχιστον τρία κράτη-μέλη για να υπάρχει επαρκής γεωγραφική κάλυψη να υπάρχει δηλαδή κινητικότητα για τους ανέργους άνω των 35. Οι προτάσεις που θα θέλαμε θα θέλαμε να έχουν ελάχιστη διάρκεια 18 μηνών. Πιστεύουμε ότι θα λάβουμε τουλάχιστον 3-4 καλές προτάσεις Και θα στηρίξουμε λοιπόν έτσι ε, αρκετά άτομα άνω των 35 για να ελέγξουν κατά πόσο μπορούν να πάνε σε άλλη χώρα για να βρουν θέσεις μαθητείας, ε, θέσεις πρακτικής εξάσκησης κτλ. Τώρα το πρόγραμμα εγγύησης για την παιδική ηλικία, για τα παιδιά, προτάθηκε από το Κοινοβούλιο ως νέα προπαρασκευαστική δράση με χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων για το 2017. Αυτή η πιλωτική δράση θεωρούμε ότι είναι συμπλήρωμα της σύστασης για την επένδυση στα παιδιά που εγκρίθηκε το 2013 που είναι σε φάση εφαρμογής με διάφορα χρηματοδοτικά μέσα στα πλαίσια της ε, ε τρεχούσης περίοδου προγραμματισμού. Υπάρχουν πέντε τομείς ε, που θέλουμε να στηρίξουμε. Τα παιδιά που κινδυνεύουν από τη φτώχεια να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, φροντίδα για τα παιδιά, αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή διατροφή μέσω των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων δράσης και προτείνουμε ο, επειδή αυτό είναι συμπλήρωμα, δεν είναι προπαρασκευή νέας νομοθεσίας, είναι περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών ε, στήριξης των παιδιών, της ανάπτυξης των παιδιών. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε η δράση αυτή να ενταχθεί στο πρόγραμμα κοινωνικής ε, ε, καινοτομίας, απασχόλησης. Θα τροποποιήσουμε λοιπόν αυτό το easy τον Ιούνιο. Δεν νομίζω ότι θα έχουν αντίρρηση τα κράτη-μέλη να υπάρξει αυτό το νέο πρόγραμμα. Αυτή η ιδέα για να γίνει μια ε, μελέτη εφικτότητας εντάσσεται πολύ καλά στο πρόγραμμα για την κοινωνική καινοτομία και την απασχόληση για να υπάρξει επαρκή κοινωνική προστασία, να καταπολεμηθεί ο αποκλεισμό και η φτώχεια. Και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλό πρόγραμμα στα πλαίσια του EASY για φέτος. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να ξεκινήσει στην αρχή του φθινοπόρου και αρχές του επόμενου έτους ε, να υπάρξει η πλήρης εφαρμογή. Ευχαριστώ Είμαι στη διάθεσή σα ε, και για ερωτήσεις για άλλα προγράμματα για τα οποία μπορεί να έχω ενημέρωση, αλλά στο βαθμό που θα την έχω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την περιεκτική παρουσίαση. Να δώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή και στους Κιώδης ε, για τον προϋπολογισμό. Ε, φυσικά όχι για το δικό του κείμενο, αλλά για τα όσα μόλις ακούσαμε τα προγράμματα αυτά. Κύριε Κλώου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή που ήρθε εδώ να μας κάνει μια παρουσίαση της πρόοδου για τα διάφορα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Είναι πολύτιμα εργαλεία ε, όλες αυτές οι νέες δραστηριότητες, νέες πολιτικές. Ε. Είχαμε την πολύ επιτυχή εφαρμογή πιλωτικών προγραμμάτων παλιότερα και ξέρω ότι καλό είναι που αυτή τη στιγμή έχουμε μια ευκαιρία να δούμε τι έχει γίνει με τα όσα έχουν ήδη εφαρμοστεί ε, τα τελευταία χρόνια καθώς προετοιμάζουμε τον προϋπολογισμό μέσα στους επόμενους ε, μήνες. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρουσίαση αυτή που είχε ζητηθεί αρχικά, όπως είπατε, από τους συντονιστές μας. Τα δύο θέματα που είδαμε σήμερα το πρωί αντικατοπτρίζουν ε, και τη ε, σημεία που ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας, ε, τους μακροχρόνια ανέργους. Η κινητικότητα των μαθητευομένων πιστεύω είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ σημαντική. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν Αυτά τα 2 εκατομμύρια για το 2007 και τα 840.000 που είπατε και τα 2,4 ε, εκατομμύρια. Πόσες χώρες πιστεύετε θα συμμετάσχουν στην ε, ε των συμμετοχών που είχαμε πέρυσι. Πόσοι πιστεύετε και πόσα άτομα συμμετείχαν τον τελευταίο χρόνο. Διότι αυτή τη στιγμή εστιαζόμαστε περισσότερο στην επαγγελματική κατάρτιση. Είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις ικανότητες του εργατικού δυναμικού για την αγορά και για τη βιομηχανία. Πόσες χώρες λοιπόν συμμετέχουν σε αυτό και στο πλαίσιο των πιλωτικών δράσεων είπατε ότι υπάρχει μια κοινοπραξία τριών κρατών μελών. Μόνο τρία. Μπορείτε να το αναλύσετε λίγο γιατί δεν το κατάλαβα πολύ καλά. Πώς γίνεται στην πραγματικότητα. Τώρα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και το πιλωτικό πρόγραμμα που σχετίζεται με αυτές και το οικοσύστημα βλέπουμε πολλές χρηματοδοτήσεις στα πανεπιστήμια μας και στον τομέα αυτό έχει τα απαραίτητα απατολίσματα. Ε, εστιαζόμαστε παρκώς ε, στο να δαπανηθούν αυτά τα χρήματα όπως πρέπει ε, και αξιολογούμε τα αποτελέσματα. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για αυτό και για το τι πρόοδο Ευχαριστώ. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστούμε. Ο Σέργιο Γκουτιέρες Πρέτο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση, την πρόσφατη ενημέρωση για το πώς προχωρούν τα προγράμματα. Είναι πολύ σημαντικές οι πιλωτικές δράσεις για να καταλάβουμε τα δύο που είναι πολύ σημαντικά, κατά τη γνώμη μου. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία Μέσω του προπολογισμού χρηματοδοτούμε προγράμματα στον κοινωνικό τομέα, στον τομέα της απασχόλησης, ε, της επαγγελματική κατάσταση, για να ενισχύσουμε τις προσπάθειες των κρατών μελών. Η ποσότητα που υποβάλλουμε εμείς για πιλωτικά προγράμματα μέσω τροπολογιών καταδεικνύει ακριβώς αυτή την αντίφαση. Από τη μία έχουμε την αρχή της επικουρικότητας, αλλά οποτεδήποτε μπορούμε ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει θέματα που ενδιαφέρουν ορισμένους συναδέλφους. Εγώ πιστεύω στην προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ λοιπόν ότι τα πιλωτικά προγράμματα ακριβώς αποδεικνύουν ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία. Αυτή ζητάμε ως Επιτροπή Απασχόλησης και στην ουσία καταδεικνύουν και τις ανεπάρκειες του κοινοτικού προϋπολογισμού. Δεν επαρκεί για να έχει την αναγκαία επίπτωση για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις που ανακύπτουν ε, στις κοινωνίες μας. Αν εξετάσουμε τα περισσότερα πιλωτικά προγράμματα που υποβάλλονται έχουν να κάνουν με τον αποκλεισμό, για να βοηθήσουμε τους ανέργους άνω των 35, την εγγύηση για τα παιδιά, ακριβώς για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια των παιδιών, των ανηλίκων είναι μια σειρά από άλλα θέματα. Η, τα start-up, ε, η ψηφιοποίηση. Προσπαθούμε να βοηθήσει λοιπόν σε όλα αυτά τα θέματα Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δείχνει επίσης πόσο είναι ανεπαρκής ο ενωσιακός προπολογισμό. Δεν καταφέρνουμε να χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά που απαιτεί η κοινωνία, που απαιτούμε εμείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση αυτά που ακούμε από την κοινωνία. Είναι πολύ καλό εργαλείο τα πιλωτικά προγράμματα αλλά αποδεικνύει απλώς σε μικρό βαθμό πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε για αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με τα εξής. Η εγγύηση για τα παιδιά. Είναι μια πρόταση που έχουμε υποβάλει εδώ και τρία χρόνια ως Επιτροπή Απασχόλησης για να καταπολεμήσουμε την ε, φτώχεια των πιο ευάλωτων που έχουν θυγεί πολύ από την οικονομική κρίση και από τις λάθος απαντήσεις, λάθος αντιδράσεις στην κρίση. Θέλουμε λοιπόν να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα η εγγύηση για τα παιδιά, ούτως ώστε να καταδειχθεί ότι και εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Επίσης η καταπολέμηση της ανεργίας. Υπάρχουν προτάσεις που είναι πολύ καλές, πολύ σωστά παρουσιασμένες. Αλλά πρέπει να επιμείνουμε, να επιμείνουμε για να καλύψουμε, ε, να αντιμετωπίσουμε όλες τις πληγές της ε, οικονομικής κρίσης. Πρέπει να κάνουμε, μια περισσότερη, να κάνουμε περισσότερη προσπάθεια, ούτω ώστε αυτή η έξοδος από την κρίση που μας δείχνουν τα μακροοικονομικά στοιχεία να σημάνει και έξοδο από την κρίση του συνόλου της κοινωνίας και των πιο ευάλωτων ε, τμήματων που έχουν μείνει στο περιθώριο της ανάκαμψης. Αυτά τα δύο πιλωτικά προγράμματα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να προχωρήσουν και να έχουν ε, την ε, μεγαλύτερη δυνατή χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Δεν έχουμε κανέναν από το Η κυρία Χάρκιν δεν είναι εδώ. Η κυρία δεν είναι εδώ, λοιπόν. Εγκούε. Ούτε. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Τζέιν Λάμπερτς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Έχω κάποιες ερωτήσεις και εγώ. Η πρώτη από αυτές αφορά την ε, επικοινωνιακή στρατηγική των πιλωτικών προγραμμάτων και παρασκευαστικών δράσεων. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και όπως είπαν και άλλοι έχουν ευρύτερε επιπτώσεις στην κοινωνία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και δεν αφορούν μόνο ε, την ελίτ και τις ε, προηγμένες ε, ομάδες, αλλά αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να δούμε τη στρατηγική μας και θα ήθελα να ασχοληθεί και η Επιτροπή μας με αυτό, εάν δηλαδή μπορούμε να βρούμε πώς να έχουμε διαρκή επικοινωνία με τους συμμετέχοντες σε αυτά τα προγράμματα. να είμαστε σε επαφή μαζί τους. Αναφέρατε την συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω περισσότερα. Να μας πείτε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μαθητεία, θα μπορούσατε να μας πείτε τι γίνεται στους επιμέρους τομείς. Για παράδειγμα, είχαμε μια έκθεση για τις πράσινες θέσεις απασχόλησης και θα πρέπει να κοιτάξουμε και την κινητικότητα μεταξύ των τομέων, εκτός από τη διασυνοριακή. Και το πώς αυτές οι δύο συνδέονται. Να δούμε δηλαδή αυτήν την τομεακή προσέγγιση, η οποία νομίζω πως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για το FDD, νομίζω δεν είναι κανείς. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ είμαι εδώ για να συζητήσουμε και έχω μια ερώτηση για την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρεις για την ακρίβεια, πολύ σύντομες. Πρώτα, η προστασία της αγοράς εργασίας, η προστασία της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για το άτομα με αναπηρία είναι πολύ βασική και πρέπει να διέπεται από κάποιες αρχές. Είμαστε μια πολιτισμένη ήπειρος και ένα κομμάτι αυτού του πολιτισμού είναι να αντιμετωπίζουμε με σεβασμό τα άτομα με αναπηρία. Μετά, η ανεργία των νέων ποια μέτρα λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω την εντύπωση πως λέμε πολλά γι' αυτό, ωστόσο νομίζω πως υπάρχουν ακόμα μεγάλα ποσοστά άνεργων νέων. Λέγονται πολλά, γίνονται λίγα. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε, θεωρώ, του ηλικιωμένου, ε, όσου ε, βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότηση. Και όχι μόνο ε, τα άτομα με αναπηρία ή με δυσκολία στην κινητικότητα. όλες τις ομάδες ανθρώπων που μπορούν να λειτουργήσουν εν είδη εφεδρικών, εφεδρικού εργατικού δυναμικού. Χρειάζεται λοιπόν να κινητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι για να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Φυσικά υπάρχουν διάφορα είδη απασχόλησης και ε, σε ορισμένους τομείς ε, τα ωφέλη δεν είναι μόνο κοινωνικά και οικονομικά, αλλά και πολλές φορές ανθρωπιστικά. Ε, με την απασχόληση αποφεύγεται η περιθωριοποίηση, η απομόνωση. Ευχαριστούμε κύριε του Γιάννη Μαρτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν συντομία, διότι δεν είμαστε παρά στην αρχή, αυτά τα πιλωτικά προγράμματα και οι σχετικέ δράσεις που μας παρουσιάστηκαν εδώ είναι γεμάτες καλές ε, προθέσεις ε, και πολύ λογικέ. Ωστόσο, υπάρχει το πρόβλημα ακόμα των μεταναστών και της κινητικότητα, Και επίσης προπολογισμοί πολύ χαμηλοί φαίνεται σαν να κάνουμε κάποιε επιφανικέ κινήσει χωρί συγκεκριμένε δράσει. Και επίση και το ερώτημα του για ποια κράτη-μέλη πρόκειται. Διότι σχηματίζει κανεί την εντύπωση ότι είναι πολύ μειωμένη εμβέλεια. Και η πρώτη αίσθηση που έχω σχηματίσει είναι ότι για άλλη μια φορά διαχειριζόμαστε περισσότερο τα αποτελέσματα τη κρίση παρά να αντιμετωπίζουμε τι πραγματικέ αιτίε που όλοι γνωρίζουμε. Τα, η λιτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σχετικά μέτρα, το κοινωνικό dumping εντός της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Τόμας Μάνου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με την αναγκαία πειθαρχία, διότι πάντα μας ρωτάνε τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν πολλά ψηφίσματα που κατεβάζουμε, πολλές δηλώσεις προθέσεων, όμως ε, πιστεύω πως πρέπει να δώσουμε αυτό που χρειάζεται, δηλαδή αποτελέσματα. Η εγγύηση για τους νέους είναι ένα υποδειγματικό ε, σύστημα, υποδειγματικό μοντέλο. Το θέμα όμως είναι να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητηθεί το θέμα της εγγύησης για τους νέους, να δημιουργηθούν ε, προϋποθέσεις, να εφαρμοστεί ε, το πρόγραμμα για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Επιτέλους ε, τα κράτη-μέλη κατάλαβαν πω μπορούν να υποφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα πως ε, και μετά θέλουν να έχουν τον έλεγχο αυτών των προγραμμάτων και αυτό είναι πολύ λογικό. Χρειάζεται λοιπόν να κοιτάξουμε επιμέρους πιλωτικά προγράμματα έτσι ώστε να πούμε στα κράτη-μέλη ότι αυτά είναι διάφορα ε, μοντέλα, συστήματα που μπορούμε να υιοθετήσουμε, να προσαρμόσουμε κατά περίπτωση γιατί εδώ βρίσκεται η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και νομίζω πως πρέπει να αλλάξει η επικοινωνιακή μας στρατηγική, διότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται σωστά. Έχουμε κάποια κονδύλια και πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά. Και πολλές φορές στην αρχή τα κράτη-μέλη ε, μπλόκαραν αυτά τα προγράμματα. Όμως πιστεύω πως ε, τώρα επιτέλους έχουν καταλάβει την σημασία τους. Έχουμε καταφέρει με αυτά τα προγράμματα να μειώσουμε την ανεργία των νέων, υπάρχουν καλές συνεργασίες, πρέπει όμως όλοι να κάνουν τη δουλειά τους, έτσι ώστε να έχουμε σωστό αποτέλεσμα. Και τώρα θα ήθελα να τονίσω και εγώ αυτό που είπε η Τζιν Λάμπερτ. Χρειάζεται επικοινωνιακή στρατηγική. Πώς θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να καταλάβουν οι πολίτες ότι εμείς ε, κάνουμε πράγματα, γίνεται δράση. Υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα τα οποία ε, δίνουν απτά αποτελέσματα. Δεν είναι απλά κάτι στο διαδίκτυο. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε ότι κάνουμε έργα και να μην πλέκουμε το εγκόμιο του εαυτού μας, αλλά να στηρίξουμε τα κρατημέλη στην προσπάθεια αυτή. Είναι πιστεύω πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό θα με ενδιαφέρε να μάθω πώς μπορούμε να το καταφέρουμε, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ποιότητα της επικοινωνίας που έχουμε, πώς μπορούμε να δώσουμε... Ε, στους πολίτες να καταλάβουν ότι υπάρχουν κονδύλια τα οποία χρησιμοποιούνται για αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό να καταλάβουν όχι μόνο οι πολίτες και τα κράτη-μέλη γενικότερα ότι τα θεσμικά όργανα είναι εκεί για να τους βοηθήσουν. Ευχαριστώ. Θα πάρω και εγώ το λόγο. Ήθελα να επανέλθω στο πρόγραμμα που σχετίζεται με τη μαθητεία, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό και πολύ επικαιρό. Έχω δύο ερωτήσεις. Αφενός ε, βάσει αυτής της δυναμικής πώς ε, ε, εφαρμόζεται τους κοινωνικούς εταίρους, πώς, πώς, γίνεται, ε, πώς τους εμπλέκεται, διότι είναι σημαντικοί συμμετέχοντες. Συχνά μιλάμε για επανεκκίνηση, ε, αναζωογόνηση του κοινωνικού διαλόγου στην Ευρώπη. Εκόντως το Ευρωπαϊκό Συνδικάτο και το Business Europe ουσιαστικά ακούω την ίδια ανάλυση, τα ίδια αιτήματα, τις ίδιες ανάγκες, οπότε ίσως εδώ έχουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να απλουστεύσει και να δει σε μια πολύ σημαντική συμφωνία για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεύτερον, το εξηγήσατε στην παρουσίασή σας, ε, ε, η χρόνη είναι πολύ μεγάλη σε άλλες χώρες. Ε, δηλαδή το ζήτημα της γλώσσας, η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας είναι κάτι σημαντικό αλλά εκεί υπάρχει επίσης κίνδυνος περιορισμού της κινητικότητας ε, των μαθητευομένων σε κατηγορίες νέων που είναι σχετικά ευνοημένοι, για να το πω έτσι. Προσπαθείτε λοιπόν να, να λάβετε υπόψη και το κοινό που είναι πιο μακριά από την απασχόληση και που βρίσκει κανείς ε, στους σημερινούς μηχανισμούς ε, επαγγελματικής ένταξης εντός Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις ε, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα έχουμε ακούσει και αυτές οι πιθανές οδοί, αλλά πρέπει να πάμε πιο πέρα ακόμα. Και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ των κέντρων εκμάθησης σε διάφορες ε, χώρες, αν αυτό σας φαίνεται δυνατό. Το θέμα είναι το εργαλείο αυτό να είναι ορατό. Ε, και να προσθέτει αξία, να αναγνωρίζεται από τους νέους ε, και να θέλουν αυτοί να συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο μαθητείας ε, διακρατικής. Το δεύτερο ερώτημα, αυτή η προβληματική που έχουμε για την ισοδυναμία των διπλωμάτων και των διαφόρων ικανοτήτων, αυτό θα χρειαστεί σε βάθος μελέτη. Και επίση έχουμε και κάποιε άλλε ιδιαιτερότητε στην Ευρώπη. Ε, και ε, μιλάμε τώρα για τι παραμεθωρίε περιοχέ. Εγώ ζω σε μια τέτοια περιοχή όπου πολλέ μικρέ και πολύ μικρέ επιχειρήσει κάνουν πραγματικέ προσπάθειε για να εκπαιδεύσουν μαθητευόμενου. Και ξέρετε ότι αυτή η εκπαίδευση είναι χρόνο, είναι χρήμα, ε, θέλει πολύ κέφι και πολύ δουλειά. Διότι είπε και ο κίνδυνο οι διπλανές χώρε να, μα, να μας βουτήξουν αυτούς τους νέους μαθητευόμενους ε, διότι α πούμε στο Λουξεμβούργο μπορεί να κερδίσουν περισσότερα ε, στο Λουξεμβούργο πούμε, μπορεί να κερδισει κανει κανείς 30-50% παραπάνω από ό,τι στη Γαλλία ένα νέο μαθητευόμενος τόσο καλύτερο για αυτόν βέβαια αλλά δεν συμφέρει αυτό του επιχειρηματίε που εκπαιδεύουν του νέου. οπότε πρέπει να δούμε κατά πόσο σε αυτά τα πιλωτικά έργα σε αυτά τα πιλωτικά προγράμματα υπάρχει η δυνατότητα να υποστηρίξουμε κάπως τις προσπάθειες αυτών των επιχειρηματιών που μπαίνουν στο παιχνίδι και που μερικές φορές ε, χάνουν όταν βλέπουν ε, οι νέοι που έχουν εκπαιδεύσει αυτοί να φεύγουν. Ενώ συχνά ο σκοπός τους ήταν να τους διατηρήσουν, να τους κρατήσουν ε, στις επιχειρήσεις τους. Κάτι άλλο που πιστεύω ότι θα χαρακτηρίσει όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια γενικότερα είναι πώς θα απλουστευθούν ε, οι αιτήσει ε, και πώς θα γίνουν πιο γρήγορα τα πράγματα και κυρίως τα χρήματα που ε, δεσμεύονται για τέτοιες δραστηριότητες να φτάνουν πραγματικά σε αυτούς που καταβάλουν τις προσπάθειες. Και ένα άλλο ερώτημα, διότι μιλήσατε για αξιοπρεπή στέγαση και κινητικότητα. Πώς ε, νοείται κατά την άποψή σας η ε, σωστή στέγαση εννοείται να είναι δωρεάν, η στέγαση και, ε, και το ταξίδι και η μεταφορά. Ξέρετε αυτά είναι κονδύλια σημαντικά για τους μαθητευόμενους και επίσης το επίπεδο αμοιβή, το επίπεδο αλλάξης της αμοιβή. Διότι καλό είναι να δίνουμε κίνητρα για την διασυνοριακή κινητικότητα, αλλά όλα εξαρτάται από το που θα πάει κανείς. Άμα πάτε σε μια χώρα με υψηλότερους ε, μισθούς ε, όπου θέλει να πάει ένας άλλος κόσμος, εντάξει, αλλά ζητήστε από νέους Γάλλους μαθητευόμενους να πάνε να κάνουν ε, μαθητεία στη Ρουμανία, δεν νομίζω ότι θα τους ελκύσει ιδιαίτερα η αμοιβή εκεί πέρα. Ευχαριστούμε. Ακούσαμε διάφορες ερωτήσεις, παρατηρήσεις πολλές ε, ήταν για εσάς και έτσι δίνουμε το λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για το ενδιαφέρον που δείχνετε και τις ερωτήσεις σας. Θα απαντήσω λοιπόν με τη σειρά που έγιναν οι ερωτήσεις. Έχουμε 4 εκατομμύρια και 800.000 επιπλέον ε, αναλήψεις υποχρεώσεων από το προηγούμενο έτος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω με ακρίβεια πόσες χώρες θα κάνουν αίτηση και πόσες θα ε, λάβουν χρηματοδότηση. Όμως ε, τα έργα αυτά θα μας βοηθήσουν να χαράξουμε νέα πολιτική που θα βασίζεται πάνω σε αυτά τα προγράμματα και τις ε, προπαρασκευαστικές δράσεις. Στοχεύουμε λοιπόν να έχουμε ας πούμε 15 κράτη-μέλη που θα καλύπτουν ε, αυτές ε, τις προτάσεις που θα απαντήσουν στην προκήρυξη και στόχος είναι να έχουμε τουλάχιστον τρία κράτη-μέλη σε μια κοινοπραξία μιας ε, παρουσίαση πρότασης. Τώρα, μπορεί πάνω από ένα κράτος μέλος να παρουσιάσει πρόταση, ιδιαίτερα αν ε, αυτή θα έχει άμεσε θετικέ επιπτώσει στην διασυνοριακή κινητικότητα και θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε δίκτυα. Όπως είπα και πριν, προσπαθούμε να εντοπίσουμε ποια είναι τα καλύτερα έργα τα οποία θα μας δώσουν τις ε, καλύτερες εφαρμόσιμες ιδέες. Έχουμε τώρα περιορισμένο προπολογισμό, ιδιαίτερα για αυτά τα πιλωτικά προγράμματα και τι προπαρασκευαστικέ δράσει. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πω πρέπει να ε, στοχεύουμε στο να δείξουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και αυτό θα γίνει κατανοώντας το σκεπτικό πίσω από κάθε πιλωτικό πρόγραμμα και προπαρασκευαστική δράση, να δούμε ποια είναι τα νέα μοντέλα που θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα εφόσον στεφθούν με επιτυχία τα προγράμματα αυτά στα κράτη-μέλη. όχι μόνο όμως ε, μέσω των ευρωπαϊκών κονδύλων, αλλά και ε, εθνικής ε, χρηματοδότησης που θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αλλά και αντιλώντας από τα διορθωτικά ταμεία. Τώρα, συμφωνώ μαζί σας, υπάρχουν πολλά πιλωτικά προγράμματα που εφάπτονται της κοινωνικής διάστασης και αυτή είναι και μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το κοινωνικό στοιχείο, δηλαδή, κάθε πολιτικής είναι Λέωνα και πιο σημαντικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κάθε πολιτική μας εξετάζεται και υπό το πρίσμα του κοινωνικού αντικτύπου. Τώρα, η συμπερίληψη των κοινωνικών εταίρων που ανέφεραν ορισμένοι συνάδελφοι, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως προτεραιότητα ε, την ε, αναβίωση του κοινωνικού μοντέλου, τη συμπερίληψη των κοινωνικών εταίρων στην χάραξη πολιτικής, στη συζήτηση. Έτσι λοιπόν, σε κάθε ε, πρόγραμμα που καταρτίζουμε και σε κάθε, κάθε μια προπαρασκευαστική δράση προσπαθούμε να συμπεριλαμβάνουμε τους κοινωνικούς εταίρους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης και εφαρμογής. Η συμμετοχή λοιπόν είναι προαπαιτούμενο και πρέπει να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, όχι μόνο να έχουν τη δυνατότητα. Υπάρχουν μάλιστα ορισμένες περιπτώσεις προγραμμάτων όπου οι κοινωνικοί εταίροι είχαν δείξει ιδιαίτερη δράση στην ανάπτυξη ε, νέων πολιτικών και νέων μοντέλων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εργαζόμαστε πολύ ε, στενά με τους κοινωνικούς εταίρους, όχι μόνο για τα πιλωτικά προγράμματα, αλλά και ε, μέσω το ΕΦΣΥ. Προωθούμε λοιπόν έναν κώδικα δεοντολογίας για τις εταιρικές σχέσεις και πέρα από την ε, υλοποίηση των προγραμμάτων έχουμε στενή συνεργασία. Τώρα, συμφωνώ μαζί σας ότι η καλή επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Προσπαθούμε δηλαδή, όπως είπα, να αναπτύξουμε νέα μέτρα, νέες μεθόδους, μοντέλα. Όμως, εάν δεν έχουμε καλή επικοινωνία, εάν δεν ενημερώνουμε, θα χάσουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Για σχεδόν όλα λοιπόν τα προγράμματα υπάρχει μια επικοινωνιακή στρατηγική που αφορά πρώτα μία στρατηγική ενημέρωση του κοινού για το τι ετοιμάζουμε, ποια είναι ε, τα προτινόμενα έργα, είναι, ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα, τι, πότε θα γίνουν προκηρύξεις και προτάσεις, ποιοι είναι οι στόχοι που θέλουμε να επιτευχθούν. Μετά δημοσιεύουμε αυτές τις πληροφορίες και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της εφαρμογής, έχει μια επιτροπή, η οποία συνεδριάζει τακτικά και τα προγράμματα κοινωνικής καινοτομίας επίσης έχουν μια τέτοια επιτροπή. Συνδυάζουμε λοιπόν αυτές τις δύο επιτροπές, γίνονται συνεδριάσεις από κοινού ε, για να συζητηθούν τα προγράμματα που εφαρμόζονται από κοινού. Και φυσικά και γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη ε, εργάζονται λίγο απομονωμένα. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να προωθήσουμε όχι μόνο ανταλλαγή γνώσεων αλλά και εμπειρίας και ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διάφορες ε, ιδέες ε, της, στην κοινή διαχείριση προγραμμάτων. Εδώ δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε καλά επίπεδα υλοποίησης, όμως ε, προσπαθούμε. Μετά, συμμετοχή. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουμε φυσικά να συμμετέχουν και να είναι δικαιούχοι των ε, προγραμμάτων μαθητείας. Και τώρα έρχομαι και στο σχόλιο ενός συναδέλφου Και θα απαντήσω λέγοντας ότι καταρχάς πρέπει να φροντίσουμε όλες οι επιχειρήσεις να έχουν ίση πρόσβαση σε αυτά τα έργα και να έχουν εξίσου καλή στήριξη. Και να διασφαλίσουμε επίσης ότι ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε προγράμματα μαθητείας, θα έχουν τη δυνατότητα μέσω αυτών να προσλάβουν νέους υπαλλήλους. Και σε ό,τι αφορά τα πλωτικά προγράμματα μαθητείας, να πω ότι θα υπάρχει πρόγραμμα γλωσσικής στήριξης, αλλά και οι μαθητευόμενοι γενικότερα θα στηρίζονται, θα μαθαίνουν πώς είναι να εργάζεσαι σε μία επιχείρηση, είτε αυτή είναι μικρή είτε είναι μεγάλη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η προσπάθεια να έχουν πρόσβαση και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτά τα προγράμματα. Τώρα, δεν έχουμε εντοπίσει συγκεκριμένους ε, τομείς ε, που είναι πάνω από άλλους. Δεν αποκλείουμε κάποιους τομείς, διότι ο στόχος μας είναι πάνω απ' όλα να γίνονται καλά προγράμματα σε όποιον ε, τομέα και αν αυτά γίνονται. Δεν, υπάρχει δηλαδή κάποιε, δεν υπάρχουν κάποιες προκαθορισμένες προτιμήσεις. Δεν αποκλείονται κάποιοι τομείς τώρα ε, για τις προβλέψεις ε, του τι θα γίνει στην αγορά εργασίας για τα άτομα με αναπηρία. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να πιέσουμε έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές πολιτικές να συμπεριλαμβάνουν ε, και τα άτομα με αναπηρία, να υπάρχει δηλαδή μη διάκριση. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς δεχόμαστε τις προτάσεις που θα συμπεριλαμβάνουν και τα άτομα με αναπηρία, που δεν θα αποκλείουν τη συμμετοχή τους. Είναι λοιπόν μία νέα αρχή που εφαρμόζουμε και ελπίζουμε να συμπεριληφθεί σε όλα τα στάδια του προπολογισμού. Τώρα, τι μέτρα έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά το 2013, μετά δηλαδή τη δημιουργία της ε, πρωτοβουλίας για τους νέους που χρηματοδοτηθήκε με 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουν γίνει διάφορα βήματα. Πέρυσι δημοσιεύτηκε η αξιολόγησή μας για την ε, εφαρμογή των ε, πρωτοβουλειών και παρατηρήσαμε ότι μειώθηκαν τα ποσοστά ανεργίας των νέων όμως αυτό το αποτέλεσμα δεν το αποδώσαμε μόνο στην ε, πρωτοβουλία αυτή για τους νέους, αλλά γενικότερα στην αλλαγή τη πολιτική που ε, έγινε μέσω ε, αυτών των νέων πολιτικών που εφάρμοσαν και τα κρατημέλη αλλά και λόγω διάφορων μακροοικονομικών παραγόντων. Η πρωτοβουλία λοιπόν για την απασχόληση των νέων στήριξε ιδιαίτερα περιοχές ε, που πλήττονται από μεγάλη ενεργεία των πάνω από 25%. Υπήρξαν λοιπόν πολλά επιλέξιμα κράτη-μέλη, πολλές επιλέξιμες περιφέρειες. Το 2015 είχαμε 15 κράτη-μέλη. Πέντε κράτη-μέλη δεν είχαν ε, περιφέρειες όπου η ενεργεία των νέων ήταν πάνω από 25%. Βλέπουμε λοιπόν ότι πραγματικά μειώνονται τα ποσοστά ενεργείας των νέων. και επομένως ο αντίκτυπος τη παρέμβασής μας εκεί ήταν πάρα πολύ θετικό. Και βέβαια στην ενδιάμεση αναθεώρηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού λάβαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια παραπάνω χρηματοδότηση για τα κράτη-μέλη που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα ανεργία των νέων. Τώρα, Έχουμε επίσης εστιάσει σε μία από τις ε, συστάσεις του κοινωνικού πακέτου 2013, για τους ηλικιωμένους δηλαδή αλλά υπάρχει και προτεραιότητα επενδυτική στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με στόχο να ενεργοποιήσει αυτό που λέμε ε, ενεργό γύρανση, να επιτρέψει δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας, να αναλάβουν θέσεις που τους ταιριάζουν, διότι ο κάθε άνθρωπος ε, μπορεί να συμμετέχει στην απασχόληση. Μπορεί να είναι χρήσιμο και θα έπρεπε. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιε δραστηριότητε που γίνονται στα κράτη-μέλη ε, και συμπεριλαμβάνουν όλε τι ε, ομάδε και του ηλικιωμένου. διάφορα μέτρα, διάφορες δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για εκείνους, όχι απαραίτητα σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Διάφορα προγράμματα λοιπόν που τους επιτρέπουν να αξιοποιούν στο μέγιστο τις δεξιότητές τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ε, απόρους, υπάρχουν κάποια κρατημέλη τα οποία επέλεξαν να μην συμμετέχουν ε, σε όλα τα προγράμματα, μόνο σε όσα ασχολούνται με την συμπερίληψη όλων των κοινωνικών ομάδων και έχουν επιλέξει να δώσουν στήριξη στις ηλικιωμένες ομάδες, στην ενεργό γύρανση και στο να βελτιωθεί η, ο, η ζωή ορισμένων ε, ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Εμείς έχουμε συζητήσει το θέμα των μεταναστών, της κινητικότητας, έχουμε όντως περιορισμένους πόρους, όμως θεωρούμε πως αυτά τα πιλωτικά προγράμματα στην καλύτερη περίπτωση θα μπορέσουν να μας δείξουν τι μοντέλα πρέπει να αναπτύξουμε. Δεν θεωρούμε φυσικά ότι τα κονδύλια που έχουμε επαρκούν για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα. Δεν αναμένουμε ε, λαμπρά αποτελέσματα σε όλη την ε, επικράτεια της Ένωσης με τόσο λίγα κονδύλια. Και συμφωνώ με τον κύριο Μαν, ήταν πολύ δύσκολο να ε, υλοποιηθεί η εγγύηση για τους νέους. Ήταν πολύ δύσκολο τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα, όμως ο αντίκτυπος είναι θετικός. Καταρχάς ε, υπάρχουν νέες πολιτικές για τους νέους που εφαρμόζονται. Ε, έχουν συσταθεί νέες εταιρικέ σχέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των πολιτικών αυτών και Άρχισε προσπάθεια μεταρρύθμισης ε, διαφόρων τομέων του δημόσιου τομέα μεταξύ άλλων. Προσπαθούν να γίνουν ε, διάφορες ε, συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε να επωφεληθούν και οι νέοι που ανήκουν σε ομάδες πιο περιθωριοποιημένες, που είναι πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς αυτούς. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες πρωτοβουλίες για τους νέους που προσπαθούν να φτάσουν σε αυτές τις ομάδες έγιναν και κάποιες ε, συστάσεις και πιστεύω εδώ έγινε η μεγάλη αλλαγή πορείας και έτσι καταφέραμε να φτάσουμε σε περισσότερους νέους. Ε, τώρα, η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Όπως σας είπα, προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε τους κοινωνικούς εταίρους στην όλη διαδικασία. Είναι ένα το κομμάτι αυτής. Και προσπαθούμε να δημοσιεύσουμε όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται από τη Γενική μας Διεύθυνση, να γίνονται συναντήσεις και διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, διοργανώνουμε συνέδρια και ούτω καθεξής. Και επίσης υπάρχουν διάφορα φόρα συνάντησης των κοινωνικών εταίρων, όπου θέμα είναι ο συντονισμός, η συνεργασία, το τι γίνεται σε επίπεδο ενωσιακό. Υπάρχει λοιπόν ε, διαρκή και συνεχόμενη επικοινωνία με του κοινωνικού εταίρου. του ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά και στην υλοποίησή του. Τώρα, αναγνώριση ε, δεξιοτήτων και πτυχίων. Σίγουρα αυτό είναι προπετούμενο για μια επιτυχή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη. Πρέπει μεταξύ εδώ να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα. Και δεν προσπαθούμε να δώσουμε προτεραιότητα σε διάφορες προτάσεις από εταιρείε που δεν ακολουθούν τους κανόνες. Προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι, να εφαρμόζονται οι κανόνες εξίσου από όλου. Αυτό το είπε και ο ομιλητής στο τέλος, αν μπορούμε δηλαδή να στηρίξουμε τις προσπάθειες όσων εφαρμόζουν τους κανόνες. Φυσικά. Πρώτα φροντίζουμε να διαπιστώνουμε ότι όντω εφαρμόζονται όλοι οι κανόνε σε όλα τα στάδια και στην υλοποίηση και έχουμε την ίδια προσέγγιση ε, σε όλου. Δεν θέλουμε λοιπόν να δείξουμε ιδιαίτερες προτιμήσεις σε όσου δεν εφαρμόζουν τους κανόνες. Και προσπαθούμε επίσης να απλουστεύσουμε τη διαδικασία ανάθεση, να γίνονται πιο γρήγορα αυτά. Ε, υπάρχουν κανονισμοί, δημοσιονομικοί κανονισμοί πρέπει να ακολουθούμε ε, και η διαδικασία επιλογής προτάσεων διαρκεί τουλάχιστον δύο μήνες αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε λοιπόν να επιταχύνουμε την διαδικασία. Δεν είναι πάντα δυνατόν αυτό. Και επίσης Προσπαθούμε όλες οι προτάσεις που αφορούν τη μαθητεία και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού να έχουν επαρκή οικονομική στήριξη, ιδιαίτερα για όσους πηγαίνουν στο εξωτερικό και φροντίζουμε λοιπόν να ε, έχουν αυτοί οι άνθρωποι αξιοπρεπή στέγαση. Προσπαθούμε λοιπόν να διασφαλίζουμε τα απαραίτητα έτσι ώστε να στηριχθεί η κινητικότητα. Νομίζω πως εδώ απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας. Αν όμως υπάρχει κάποια επιπλέον ερώτηση, με τα χαρά την απαντήσω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ε, έγιναν πολλές ερωτήσεις, αλλά δώσατε και πολλές απαντήσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε μία ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις. Τώρα, χρονοδιάγραμμα. Για την έκθεση για το γενικό Προϋπολογισμό με τα διάφορα στοιχεία, τροπολογίες μέχρι τις 25 Απριλίου. Συγγνώμη, τις προτάσεις για πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές ενέργειες. Θα λάβετε το χρονοδιάγραμμα, το πλήρες χρονοδιάγραμμα μέσω ε, mail γιατί αναφέρονται μια σειρά από ημερομηνίε, αλλά δεν θέλω τώρα να τις ε, αναφέρω μία-μία εδώ. Να ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ ε, κύριε Σούκοβα για τις απαντήσεις σας. Το επόμενο θέμα λοιπόν έχουμε τώρα στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της Ένωσης. Και η συγκεκριά μας είναι η κυρία Γκονθάλεφ Πένιας. Παρακαλώ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας. Είναι έκθεση πρωτοβουλία της Επιτροπής Γυναικών. Έχουμε γνωμοδότηση εμείς η ΕΜΠΛΕ. Θέλουμε να συνδυάσουμε το διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα αυτά συμπίπτουν ε, και με τις ε, προτάσεις ε, της Επιτροπής για νομικά θέματα και θεμάτων των γυναικών των Ηνωμένων Εθνών όσο και τη δική μας πρόταση για την 8η Μαρτίου είναι λοιπόν ένα θέμα στη διεθνή και ευρωπαϊκή επικαιρότητα. Υπάρχουν πολλά εμπόδια για την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των γυναικών, είναι διαφορετικά. Βέβαια είναι κάπως διαφορετική η κατάσταση στον ιδιωτικό από το δημόσιο τομέα, αλλά πρέπει να αναλύσουμε γιατί υπάρχουν αυτοί οι φραγμοί για να επιχειρήσουμε να καταλάβουμε τα κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά στοιχεία που είναι διασυνδεδεμένα και που έχουν ως αποτέλεσμα την ε, διαιώνιση αυτής της ανισότητας. Αυτό προσπαθεί να κάνει αυτή η γνωμοδότηση θέτει οχτώ ζητήματα που νομίζω ότι είναι θεμελιώδη για να επιτύχουμε λοιπόν αυτή την οικονομική βελτίωση των γυναικών στο δημόσιο και, οικονομικό τομέα, και ιδιωτικό τομέα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να υπάρχει ίση αμοιβή για ίση εργασία για να υπάρχει οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Δεύτερον, να καταπολεμήσουμε τι πιο επισφαλεί μορφέ απασχόληση που κυρίω στείλουν τι γυναίκε και που έχουν ω επίπτωση αυτή τη διαφορά στου μισθού και τι συντάξει και έχουν να κάνουν πολύ με, την, ε, με τις άτυπες μορφές εργασίας, τον εθελοντισμό και τη μερική εργασία. Επίσης πρέπει να σταματήσει αυτός ο διαχωρισμός σε επαγγέλματα που κάνουν οι άνδρες και οι γυναίκες, να μπορέσουν να συμμετάσχουν πλήρως οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, να έχουν πλήρη κατάρτιση και να υπάρχει κοινή ευθύνη για τις οικιακές εργασίες και τη φροντίδα των μελών της οικογένειας. Κάτι άλλο. Στο 4 αναφέρω ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ούτως ώστε οι εργασίες που και στο παρελθόν παραδοσιακά και τώρα που κάνουν κυρίως οι γυναίκες, όπως για παράδειγμα οι οικιακές εργασίες, η φροντίδα μελών της οικογένειας, αυτά να μην, είναι, ε, να μην θεωρούνται μικρότερες αξίες και να μην ε, φέρουν στίγμα. Πρέπει επίσης να μην υπάρχουν διακρίσεις στην επιλογή και την προαγωγή των γυναικών και στους δύο τομείς να προχωρήσει η οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών και να διασφαλίσουμε ηγετικέ θέσεις των γυναικών στα όργανα στον οικονομικό και πολιτικό τομέα όπου λαμβάνονται αποφάσεις, να ενισχυθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να υπάρξουν περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις. Και τέλος, δεν είναι δυνατόν να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών εάν δεν ε, προωθήσουμε νοοτροπίες κοινή ευθύνη για τις οικιακές εργασίες. Γιατί αυτό είναι ένας από τους διαφορετικού λόγους των ανισοτήτων. Οι τροπολογίες μου θα επιχειρήσουν να διευρύνουν την κοινωνική πλευρά, την οικονομική και κοινωνική, για να ε, βελτιωθεί λοιπόν η κατάσταση των γυναικών και στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, συμβολή των διαφόρων σκιωδών και άλλων μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ λέει και ο Πρόεδρος για το ΕΛΚ. Η κυρία Σοφία Γριμπέο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα μιλήσω αγγλικά αυτή τη φορά διότι αντικαθιστώ την Ανιέσκα Καλόφσκα σκιώδη του ΕΛΚΑ Συγγνώμη δεν μπορώ λέει, να προφέρω καλά το όνομά της Ανιέσκα η οποία ζητά συγγνώμη που δεν μπόρεσε να βρίσκεται στη σημερινή συνάντηση. Μου ζήτησε να σας παρουσιάσω τη θέση του ΕΛΚ όσον αφορά τη γνωμοδότηση για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αλλαγές που θέλει να ε, προσθεθούν. Η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών είναι ζήτημα κλειδί τόσο για τις προσωπικές ε, ζωές των γυναικών και την ευημερία τους, καθώς και για την ανάπτυξη ε, της ευρωπαϊκής οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε σημαντικές εξελίξεις στον τομέα αυτών. Στην τελευταία σύνοδο της Επιτροπής των Εθνών για την κατάσταση των γυναικών αντιμετωπίστηκε η ενδυνάμωση των γυναικών ως παγκόσμια πρόκληση και ο δικός χάρτης ε, για την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ε, ζωής προετοιμάζει διάφορες νομοθετικές και μη λύσεις για τον τομέα αυτών. Ε, το Κοινοβούλιο λοιπόν και η Επιτροπή ΕΜΠΛΑ πρέπει οπωσδήποτε να θέσουν σαφείς στόχους για την ενδυνάμωση των γυναικών και να εστιαστούν στα όσα είναι εφικτό να επιτευχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά το περιεχόμενο της γνωμοδότησης, το ΕΛΚ θα ήθελε πρώτα απ' όλα να επισημάνει ότι η ισότητα των φίλων και η ενδυνάμωση των γυναικών παρουσιάζουν πολλά ωφέλη. Πρέπει να δείξουμε ότι δεν πρόκειται για ένα παράπλευρο ζήτημα, ούτε μια πρόκληση που αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά μια οικονομική ευκαιρία που δίνει τη δυνατότητα ε, για περισσότερη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς. Επίσης, η τη ηγετρία θέλει να εστιαστεί στο πόσο αναγκαίο είναι να εφαρμοστούν σωστά οι νομοθεσίες για την κατάρριξη της διακριτικής μεταχείρισης στην απασχόληση. Υπάρχει μια τάση να προτείνεται νέα νομοθεσία διαρκώς, η οποία όμως δεν πρόκειται να βοηθήσει αν δεν ασκηθεί και δεν εφαρμοστεί πλήρως. Τρίτον, επειδή πρόκειται για γνωμοδότηση της ΕΜΠΛ, η Σκιώδης θα ήθελε ε, να προβάλλουμε το ζήτημα των οικιακών βοηθών η διευκόλυνση της απασχόλησής τους και η πρόθεση ευέλικτων λύσεων σε αυτό το τομέα είναι κάτι πολύ σημαντικό ώστε να καταπολεμήσουμε την αδήλωτη εργασία αλλά και να βελτιώσουμε την ισορροπία ε, επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αυτών των ανθρώπων. Η Σκιώδης ε, ελπίζει ότι θα υπάρξει καλή συνεργασία με τους λοιπούς Σκιώδης και, ε, ώστε να καταλήξουμε σε σωστά αποτελέσματα με βελτίωση της κατάστασης των γυναικών. Ευχαριστούμε ε, για τους σοσιαλιστές Άγνες ε, ε, Γιόγκερος. Ευχαριστώ και εγώ εκπροσωπώ τη μία Πέτρα η οποία δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ σήμερα και μου ζήτησε να διαβάσω τις σημειώσεις της. Για μας το σημαντικό είναι αυτό που λέει η έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ισότητας των Φύλων, ότι ε, μια βελτίωση της ισότητας θα προσθέσει 10,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέχρι το 2050 που θα αυξήσει το κατακεφαλήν ΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 6 ε, ποσοστία σημεία. Αυτό αποδεικνύει πόσο σημαντικές είναι οι γυναίκες για τις αγορές εργασίας. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό ε, σε αυτή την περίπτωση όταν εργάζονται και οι δύο γονείς είναι η εξισορρόπηση μεταξύ προσωπικής ε, και επαγγελματικής ζωής. Αν δεν υπάρχουν ε, υπηρεσίες επαρκής περιπτήσης των φροντίδας των παιδιών, οι γυναίκες δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι και να εργαστούν. Οπότε το πρώτο ζήτημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτή η εξισορρόπηση της οικογενειακής και ε, επαγγελματική ζωής, δηλαδή οι γυναίκες να μπορούν να έχουν μια ισορροπημένη οικογενειακή ζωή. Η άδεια μητρότητα θα πρέπει να διασφαλίζεται για όλες τις γυναίκες. Το δεύτερο ζήτημα, κάτι αναγκαίο για να μπουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, μια νέα μορφή εκπαίδευσής τους, ε, διαρκούς ε, διαβίου εκπαίδευσης ε, μέσω εμπειρίας, κατάρτισης, επικαιροποίησης των, ε, αναβάθμισης των ικανοτήτων στον ψηφιακό κόσμο, απαραίτητο για να βρει κανεί δουλειά σήμερα και ακόμα και αν δεν δουλεύουν, ε, ξέρετε, κάποιοι μπροστά σε υπολογιστή, ορισμένα επαγγελμάτα απαιτούνται κάποιε ψηφιακέ δεξιότητε. Είτε παραγγέλνει κανεί νέα προϊόντα, είτε ε, συμπληρώνει τις ώρες εργασίας του. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε οι γυναίκες να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε όλους τους τομείς. Οι γυναίκες είναι αναγκαίες ε, ε, στις θετικές επιστήμες, στη φυσική, στα μαθηματικά, όπου ο κόσμος είναι κυρίως, ε, όπου οι άνθρωποι είναι κυρίως άνδρες. Αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει ως νοοτροπία. Χρειάζεται και περαιτέρω εκπαίδευση ώστε να ενθαρρύνουμε περισσότερες γυναίκες να φοιτήσουν σε αυτούς τους τομείς. Το τρίτο σημείο που μου φαίνεται σημαντικό είναι η ένταξη των γυναικών σε διάφορα επίπεδα διαφορετικής φύσης. Αναγνώριση δεξιοτήτων και άτυπων και τυπικών δεξιοτήτων. Αυτά είναι όλο και πιο σημαντικά ε, στις νέες αγορές εργασίας. Ο κόσμος ε, κάνει εθελοντισμό, μαθαίνει πολλά μέσα αυτού. Μαθαίνει πολλά και για τις ψηφιακές τεχνολογίες. Οπότε δεν μπορούμε να ε, θεωρούμε ότι το να παρακολουθεί κανείς μαθήματα σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα σχολείο αρκεί. Ένα τέταρτο ζήτημα είναι οι γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστες. Χρειάζονται ενθάρρυνση, συμβουλευτική υποστηρίξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Πρέπει πιστεύω να υποστηρίξουμε την πορεία τους, η οποία είναι τόσο δύσκολη και τόσο μακροχρόνια. Και τέλος, ε, ισότητα στο χώρο εργασίας. είναι κάτι για το οποίο αγωνιζόμαστε εδώ και πολλές δεκαετίες. Ε, ε, οι πιστολογικέ διαφορέ, ε, το πιστολογικό χάσμα, το συνταξιδοτικό χάσμα είναι γνωστό σε πολλέ γυναίκε, σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Η αξιοπρεπή αμοιβή λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να θέσουμε ρητά ω στόχο και με διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επενδύσει έτσι πολύ αποτελεσματικά και δεν αναφέρομαι μόνο στο οικονομικό πρέπει να γίνει αυτή η επένδυση ε, υποστηρίζοντας γυναίκες επιχειρηματίες ε, στις νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω των διαφόρων ταμείων ώστε να μπορούν οι γυναίκες να, να γίνουν επιχειρηματίες με πιο ευέλικτο και λιγότερο γραφειοκρατικό τρόπο. Ο κύριος Κέρινγκε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και για αυτό το πολύ ενδιαφέρον ε, θέμα για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η ισότητα για μένα είναι ένας πολύ επικίνδυνο όρος. Γιατί ε, υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Και αν δεν ληφθούν αυτές οι διαφορές υπόψη, τότε ε, κινδυνεύουμε ε, να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερες ανισότητες. Από, από αυτό ε, λείπει η ομάδα των, των γυναικών που είναι μητέρες. Οι μητέρες δίνουν πάρα πολλά στην κοινωνία, δεν πληρώνονται γι' αυτό. Στη Γερμανία μάλιστα πολλές μητέρες φροντίζουν και παιδιά άλλων. Όμως αυτό δεν αμείβεται και πολλές φορές στους παιδικούς ε, σταθμούς φροντίζονται ε, παιδιά και πληρώνουν γι' αυτό. Ε, κάποια οικογένεια πληρώνει στους ε, παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά της, όμως η μητέρα δεν πληρώνεται που φροντίζει τα παιδιά της στο σπίτι. μετά υπάρχουν άλλα θέματα, η άδεια μητρότητας για παράδειγμα, που πολλές φορές δεν αναγνωρίζεται. Και σίγουρα υπάρχουν και άλλα θέματα, για παράδειγμα στις ε, διακοπές. Όταν, όταν πάμε ε, διακοπές ε, φροντίζουμε και εκεί τα παιδιά μας. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως και οι μητέρες θα πρέπει να έχουν άδεια από αυτές τους, τις δουλειές, από την ιδιότητα της μητέρας. Υπάρχουν πάρα πολλές ανισότητες λοιπόν οι οποίες είναι εις βάρος ε, της μητέρας και υπάρχουν, ε, υπάρχει άνηση αντιμετώπιση ε, σε αυτούς που δεν έχουν παιδιά. Υπάρχουν δηλαδή πολλές φορές διαφορές της τάξης του 40% οικονομικού χαρακτήρα ανάμεσα στα άτομα που δεν έχουν παιδιά και στους γονείς. Όταν κάποιος άτεκνος, ε, χρησιμοποιεί το επιχείρημα «Ναι, ωραία, και τι να κάνουμε, εσύ γιατί έκανες παιδιά αφού δεν μπορούσες να επομιστείς το κόστος». Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Ε, μετά, ακούσαμε και το άλλο, ότι όταν ε, δουλεύουν και οι δύο γονείς τι γίνεται. Ναι, θα πρέπει επιτέλους να αναγνωριστούν ε, και οι προσφορές των γυναικών, η δουλειά των γυναικών που είναι μητέρες και να έχουν και το δικαίωμα για άδεια. Υπάρχει λοιπόν μονόπλευρη στήριξη από το κράτος στους γονείς και πιστεύω πως πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης. Χρειάζεται οι γονείς να έχουν την ελευθερία της επιλογής, ε, του να επιλέξουν δηλαδή να κρατήσουν ένα ποσό και να μείνουν στο σπίτι να φροντίσουν τα παιδιά τους ή να ε, δώσουν τα παιδιά τους ε, σε παιδικό σταθμό ας πούμε. Χρειάζονται κέντρα για την οικογένεια που θα παρέχουν βοήθεια κάθε είδους, που θα έχουν ευέλικτα ωράρια. Χρειάζεται ευέλικτη στήριξη στους γονείς, διότι πιστέψτε με η οικονομία με αυτόν τον τρόπο θα γίνει πιο παραγωγική, θα αυξηθεί η ικανοποίηση πίση στο χώρο εργασίας και υπάρχει και ένας ε, νέος όρος που συνδυάζει την ιδιότητα της ε, μητέρας και του επιχειρηματία. Και εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε την ειδική, ε, το ειδικό βάρος που έχουν οι μητέρε. Ε, το να θεωρούμε ότι όταν μια γυναίκα μεγαλώνει παιδί ε, δεν συμμετέχει στην αγορά εργασίας είναι πιστεύω ε, λάθος. Ακούμε ότι χάνει την επαφή με την αγορά εργασίας, ότι πρέπει να προφτάσει τις εξελίξεις. Όμως εγώ θα ήθελα να ζητήσω να σκεφτούμε αλλιώ τα πράγματα, να υπάρχει ένας μισθό που θα παίρνει η μητέρα που ανατρέφει τα παιδιά της, ε, να αλλάξει το σύστημα με τους ε, παιδικούς σταθμούς έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και αυτό το μισθολογικό χάσμα και το συνταξιδοτικό χάσμα ανάμεσα στους άντρες και γυναίκες. Είναι άδικη η, ε, μεταχείριση της κοινωνίας τους άτεκνους και σε όσους έχουν παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν η ισότητα στο μισθό πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους γονείς. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Σελίμοβιτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα αρχίσω ευχαριστώντας το, την εισηγήτρια για αυτή τη γνωμοδότηση. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό σχέδιο γνωμοδότησης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, το 76% των Ευρωπαίων θεωρούν πως πρέπει να αντιμετωπιστεί η ανισότητα ανδρών και γυναικών και να γίνει μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης, εξίσου μεγάλο ποσοστό θεωρεί πως πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η ανισότητα ανδρών και γυναικών έτσι ώστε να ε, γίνει πιο δίκαιη η κοινωνία μας. Οι πολίτες λοιπόν βλέπουμε ότι έχουν, παρέχουν ευρύτατη στήριξη σε αυτό το θέμα. Και πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια πρόοδο, έχει γίνει βήμα-βήμα αυτή η, πρόεδρος, η πρόοδος και πρέπει να συνεχίσει έτσι έστει ώστε να υπάρξει ισότητα. Οι ίσες ευκαιρίες ε, όμως δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν και στον τομέα της απασχόλησης. Εδώ η πρόοδος είναι αργή. Ε, απέχουμε πολύ από το να υπάρχει ισότητα στις συντάξεις, στη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικέ θέσεις, ε, στις οικονομικές απολαύσεις κτλ. Για παράδειγμα, η ισότητα στις αμοιβές αρνητών και γυναικών ε, υπάρχει μόνο στο 17,4% της επικράτειας της Ένωσης. Όπως όμως και αν μετρήσουμε αυτά τα νούμερα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το 39% ε, και αυτό το ποσοστό αφορά την ανισότητα στις ε, συντάξεις ανδρών και γυναικών. Μετά, οι ηγετικές θέσεις κάτω από το 4% των ε, θέσεων, των υψηλών θέσεων στις επιχειρήσεις ανήκουν σε γυναίκες. Οι γυναίκες εργάζονται αμυστή κάνοντα οικιακέ εργασίε χωρί να αναγνωρίζεται αυτή η εργασία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξουμε την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Είναι μάλιστα προαπαιτούμενο έτσι ώστε να λάβουν οι γυναίκε τα πράγματα στα χέρια του, να έχουν ελευθερία επιλογών έτσι ώστε να συνεισφέρουν περισσότερο στην ε, κοινωνία. Πρέπει να αναγνωριστεί λοιπόν το έργο των γυναικών για να ε, τονωθεί και η οικονομία και η ανταγωνιστικότητα. Ε, και του τουλεχθέντος θεωρώ πως η πρόταση είναι αρκετά καλή. Θα ήθελα όμως να κάνω και μερικά σχόλια από το κειμένου έτσι ώστε να ε, δοθεί και η δική μας διάσταση. Για την παράγραφο 2 θεωρώ πως πρέπει να ε, έχει πιο φιλόδοξη διατύπωση έτσι ώστε να προωθήσει την ευημερία των γυναικών. Γιατί έτσι όπως αναφέρεται είναι πολύ υποκειμενικό το πώς θα ερμηνευτεί. Χρειάζεται λοιπόν να προωθεί η ισότητα ανδρών και γυναικών μια και η ισότητα εξάλλου είναι μία από τις θεμελιώδεις ε, αρχές ε, των συνθήκων. Επίσης, στην παράγραφο αυτή δεν βλέπω κάποια θετική διατύπωση που να αφορά τις ευκαιρίες ε, και την ευελιξία της αγοράς εργασίας. Και εμείς ως φιλελεύθεροι ε, ανησυχούμε για την έλλειψη ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Μετά, οι γυναίκες επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις και χρειάζονται λοιπόν περισσότερες δράσεις έτσι ώστε να προωθήσουν την καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την κατάρτιση, ε, την πρόσβαση σε δίκτυα επιχειρηματιών και την συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την γνωμοδότησή τη και να πω πως θα υποβάλουμε και τις δικές μας τροπολογίες, ε, οι οποίες ε, θα αντιτοπυρίζουν αυτά που μόλις ε, σα είπα και θα δείχνουν τη θέση των φιλελεύθερων. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σντανόκα, για τους πράσινους. Αντικαθιστώ τη Μόνικα Βάνα που είναι η σκιώδης μας, δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα. Και εκ μέρου τη λοιπόν, καταρχά ευχαριστώ την κυρία Γκονθάλεφ Πένιαθ για το σχέδιο γνωμοδότηση. Συμφωνούμε με την προσέγγιση τη σε γενικέ γραμμές. Θέλουμε όμως να ενισχύσουμε ορισμένα σημεία, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της ομάδας μας, ότι η βελτίωση της οικονομικής θέσης των γυναικών είναι βασικό στοιχείο για την ισότητα των φύλων. Γι' αυτό θα υποβάλουμε μία τροπολογία που τονίζει τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και τονίζει τη σημασία της άδειας μητρότητας και πατρότητας. Ξέρουμε ότι η Επιτροπή επίσης θα υποβάλει μια νέα πρόταση οδηγίας για το θέμα αυτό. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε τις ολέθρες επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας ε, για την ε, οικονομική κατάσταση των γυναικών. Ξέρω ότι δεν συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες από αυτού, αλλά η θέση μας ε, είναι ιδιαίτερα αρνητική έναντι αυτών των μέτρων λιτότητας. Επίσης τονίζουμε ε, την ε, μεγάλη σημασία των δημοσίων υπηρεσιών, των κοινοφελών υπηρεσιών. Αυτές είναι οι απόψεις που θα προβάλλουμε μέσω τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ. ΙΕΝΕΦ, ο κύριος Μαρτάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί βλέπω ότι έχετε κάποια καθυστέρηση στις ε, στις εργασίες μας. Ναι. Βελτίωση της θέσης των γυναικών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς θεωρούμε ότι 70 με 80% των γυναικών όχι μόνο είναι υποχρεωμένες να εργαστούν σε αυτή την ε, καταναλωτική κοινωνία, γιατί δυστυχώς σε αυτή την κοινωνία χρειάζονται δύο μισθοί σε ένα νοικοκυριό για να μπορέσει να, μπορέσει να ζήσει κανείς αξιοπρεπώς. Άρα είναι υποχρεωμένε και ακόμη χειρότερο. Θεωρούμε ότι 70 έως 80% των γυναικών, δεν μιλάω για το 20% που είναι θαυμάσιες, εξαιρετικέ και τα πάνε μια χαρά, όχι μόνο είναι υποχρεωμένες, αλλά είναι αντικείμενο εκμετάλλευση αυτές οι γυναίκες. Με μερική απασχόληση, ιδιαίτερα στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, σε εταιρείε καθαρισμού, όπου τους δίνουν πενταροδεκάρες, 600-700 ευρώ το μήνα και ακόμη χειρότερα. Δεν έχουν ακόμη δυνατότητα να ορίσουν πότε θα εργαστούν. Τις υποχρεώνουν να πάνε να εργαστούν. Όποτε θέλουν εκείνοι, τις εκμεταλλεύονται και τη Δευτέρα πρωί τους λένε «Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα θα δουλέψεις τότε και τότε». Άρα δεν μπορούν να οργανώσουν τη ζωή τους, δεν μπορούν να οργανώσουν το πώς θα φροντίσουν για τη ζωή τους, για τα παιδιά τους. Όλα αυτά είναι απολύτως αδύνατα. Όλες μας οι τροπολογίες θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ωραία, ακούσαμε τους διάφορους σκιώδεις. Τώρα κλείνω το κατάλογο των συναδέλφων που θέλουν να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ, δύο λεπτά ή ο καθένας. Ε, Σοφία Ριμπέιγο. Θα είμαι πολύ σύντομη. ορισμένα σημεία που πιστεύω ότι πρέπει να προσθεθούν στην ε, έκθεση. Πρώτα, λόγω των τάσεων στην αγορά εργασίας όπως προβλέπουμε ότι θα ε, υπάρξουν στο εγγύς που έχουν να κάνουν με την ε, επιστήμη, την τεχνολογία και την ανεπάρκεια της κατάρτισης των γενικών σε αυτό το τομέα κάτι το οποίο δυστυχώς και περίεργα δεν συμβαίνει στην Ευρώπη, στην Πορτογαλία αλλά συμβαίνει στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολλά για την εκπαίδευση των νέων γυναικών και των κοριτσιών στους τομείς αυτούς. Ιδιαίτερα για την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι θα μπορούσαμε βράχη και μέσω πρόθεσμα να αποφύγουμε αυτό το τεράστιο χάσμα για τους μισθούς. Όλα αυτά τα θέματα μητρότητας, πατρότητας και συνδυασμού της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τα δικαιώματα των πατέρων, των ανδρών Πρέπει οπωσδήποτε να ενισχύσουμε και τη δική τους ε, θέση και να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να χορηγούν και άδειες πατρότητας. Και να υπάρχουν ε, λοιπόν καθεστώτα απασχόλησης που θα επιτρέπουν ελεύθερα στα ζευγάρια να αποφασίσουν ποιος θα ασχοληθεί με το νεογέννητο ή για παράδειγμα με ένα ε, ανήλικο που έχουν υιοθετήσει. Δεν θα έπρεπε λοιπόν ε, τη φροντίδα για τα παιδιά να την ε, αναλαμβάνουν αποκλειστικά γυναίκες. Και εδώ πρέπει να υπάρχει ισότητα των φίλων. Όλοι θα έπρεπε να συμβάλλουν στην ανατροφή των παιδιών, όλοι θα έπρεπε να έχουν επαγγελματική δραστηριότητα. Τώρα τα ωράρια. Τρίτο σημείο. Τα ωράρια πρέπει να είναι πιο ευέλικτα για να μπορούν και οι μητέρες και οι πατέρες να είναι κοντά στα παιδιά. Ξέρουμε ότι τώρα ε, κυρίως ασχολούνται οι μητέρες και αυτό ε, δημιουργεί προβλήματα στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Και δεν μπορούν λοιπόν να συνδυάσουν ε, τη φροντίδα αυτή με την δουλειά τους. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ελαστικά ωράρια, πρέπει να υπάρχουν βρεφονιπιακοί σταθμοί, για να συμπληρώνουν τις ώρες ε, ε, όπου τα παιδιά είναι στο σχολείο, ούτω ώστε οι γονείς ακριβώς ε, που δεν μπορούν στις 4 να πάνε να μαζέψουν τα παιδιά, να μπορούν να πάνε αργότερα. Επίσης πρέπει να αναγνωριστεί η απασχόληση εντός της οικογένειας, όχι μόνο για την ανατροφή των παιδιών, αλλά και για τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Πρέπει να αναγνωριστεί αυτή η προσφορά. Είναι απασχόληση και πρέπει να υπάρχουν δύο δυνατότητες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι για να γίνει αυτή η ανατροφή, να γίνει αυτή η φροντίδα, χρειάζονται ορισμένε ικανότητε, ορισμένα προσόντα. Πρέπει να αναγνωριστούν αυτά τα προσόντα. Ιδιαίτερα για όσου ασχολούνται με πολύ μικρά παιδιά και ηλικιωμένου. Και επίση πρέπει να υπάρχουν και κοινωνικέ ε, παροχέ για τα άτομα αυτά. Να μην θίγεται ε, η υγεία τους Ευχαριστώ η κυρία Γκουτιέρεθ Πριέτο. Ο κύριος Γκουτιέρεθ Πριέτο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό που συζητάμε για την βελτίωση της κατάστασης των γυναικών. Πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε σημασία στις αξίες που θέλουμε να προωθήσουμε. Γιατί υπάρχει ένα προπατορικό αμάρτημα δεν έχει, έχουν δημιουργήσει οι κοινωνίες μας τη δυνατότητα για να μπορούν να πάρουν οι γυναίκες τη θέση που τους ανήκει. Και ακούμε ότι όλο και περισσότερο νέοι πιστεύουν σε φαλοκρατικά πρότυπα και προκαταλήψεις που εδώ και δεκαετίες προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από τη ρίζα του. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της βίας, ε, της ενδοοικογενειακής βίας και ιδιαίτερα και η παρενόχληση στον τόπο εργασίας. Γιατί υπάρχουν προβλήματα και στο εργασιακό περιβάλλον. Πρέπει να τα εκριζώσουμε. Μόνο έτσι θα βελτιώσουμε την κατάσταση των γυναικών. Χρειαζόμαστε λοιπόν και νόμους καλύτερους και μεγαλύτερους προϋπολογισμούς. Επίσης, Πρέπει να ενισχύσουμε ε, όλα τα θέματα για, την, ε, για τον συνδυασμό της προσωπικής και οικογενειακής από τη μία και επαγγελματικής ζωής. Πρέπει να αλλάξουν τα ωράρια. Ε, υπάρχουν μελέτες που λένε ότι και για τους άνδρες και για τις γυναίκες μειωμένα ωράρια βοηθούν αυτόν τον συνδυασμό. Βελτιώνουν την παραγωγικότητά μας, μας κάνουν και οικονομικά πιο επωφελείς για την κοινωνία και για την οικογένειά μας. Και φυσικά και οι άδειε μητρότητα και πατρότητα δεν είναι διακοπέ, είναι δικαίωμα. Είναι δικαίωμα για να είναι κανεί υπεύθυνο για την ανατροφή των παιδιών του. Και γιατί έχουν δικαίωμα και τα παιδιά να τα ανατρέφουν οι γονεί του. Ορισμένοι λένε, ορισμένα πράγματα ε, τα αντιμετωπίζουν με ελαφρότητα. Ορισμένοι λένε ότι ορισμένοι γονείς στην ουσία, ορισμένα ζευγάρια, είναι εργοστάσιο κατασκευή παιδιών. Αυτά δεν είναι σωστά. Πρέπει οι γονεί να μπορούν να ανατρέφουν τα παιδιά του. Θέλουμε να έχουμε ένα τέτοιο κοινωνικό πρότυπο. Θέλουμε να το επεκτείνουμε και σε άλλα μέρη του κόσμου. Άρα, πρώτα απ' όλα, να αναγνωρίσουμε ότι είναι ανεπαρκή οι άδειε μητρότητα, όπω τι έχουμε τώρα. Πρέπει να ε, αμείβονται 100% και πρέπει να προωθήσουμε και τι άδειε πατρότητα. Να είναι υποχρεωτικέ επαρκή σε χρόνο και επίση αμοιβόμενε. Με ανησυχούν αυτά τα χάσματα που έχουμε τώρα, αλλά με ανησυχεί περισσότερο το χάσμα στο μέλλον, λόγω του ψηφιακού κόσμου. Τις τελευταίες δεκαετίες δεν καταφέραμε να μειώσουμε την ανισότητα αυτά. Άρα προσθέτονται, προστίθενται δεκαετίες και δεκαετίες και τώρα με αυτή την ψηφιοποίηση μπορεί να επιδεινωθεί ακόμη η κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανισότητα αυτή που θα προκύψει λόγω της ψηφιακής οικονομίας. Κατά λίγο, Πρόεδρε. Και να αναφερθούμε και στην ε, διπλή διάκριση για τις γυναίκες που είναι και πρόσφυγες ή μετανάστριες ή που ζουν στην Ήπεθρο. Αυτές υφίστανται διπλή διάκριση. Δεν είναι λοιπόν μόνο θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, αλλά και οικονομικής αποδοτικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Εντουά ήταν δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα κάνω και λιγότερο. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά. Μερικές σκέψεις. Και εγώ είμαι νέος πατέρας. Μόλι έγινα πατέρας και πήγα στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν απέκτησα το γιο μου για να πάρω άδεια πατρότητας και μου είπαν δεν υπάρχει. Ε, η αξιοπιστία ενός ερετού είναι κατά πόσο αυτό που απαιτεί από του άλλου εφαρμόζεται στον ίδιο. Αυτή είναι μια πρώτη μου παρατήρηση. Επίση, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει απόλυτη ε, οικονομική χειραφέτηση χωρί ε, ε, κοινωνική χειραφέτηση. Πρέπει να σπάσουμε τα ταμπού, τα κλισέ. Αυτό περνάει από την εκπαίδευση. Ποιο εδώ ή αλλού δεν έχει αναρτηθεί κάτι τέτοιο όταν βρήκε δουλειά. Το κατά πόσο θα μπορέσει να συμφιλειώσει οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Ο ε, άνδρας αυτό το ερώτημα δεν τίθεται. Ωστόσο είναι ένα ζήτημα, ένα ερώτημα που τίθεται σε γυναίκες σε κάθε συνέντευξη. Ε, τα περίεργα ωράρια είναι δύσκολα, ε, ε περίεργες ώρες συνεδριάσεων, ε, τίθεται και το ζήτημα της, διφτής, της διπλής ημέρας εργασίας και μετά διαρκώς απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία ε, επαγγελματική την οποία, η οποία απορρίπτεται στον κοινωνικό τομέα. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, να είμαστε ανταγωνιστικοί ε, και αυτό απαιτεί να κάνουμε συνεδριά στις 6 το απόγευμα. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά ωφέλιμο, έχει νόημα οικονομικά για μια επιχείρηση. Οπότε εγώ συμφωνώ. Πρέπει να υπογραμμίσουμε και έντονα όλα αυτά τα θέματα και ευχαριστούμε για τη δουλειά που έχει γίνει, αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει οικονομική ενδυνάμωση και χειραφέτηση χωρί πολιτιστική και κοινωνική χειραφέτηση. Ευχαριστώ να αφήσω την εισηγήτρια την κυρία Κονζάλε Πένια να μας πει κάποια τελευταία λόγια. Δύο λεπτά το πολύ παρακαλώ. Sí, perdón. Eh, <laughs> bueno, muchas gracias a, a todos y a todas por, por las aportaciones. Creo que hay muy buenos mimbres que, que todas las, las aportaciones. Ευχαριστώ πολύ για όλα όσα είπατε όλοι. Νομίζω ότι όλες οι παρεμβάσεις πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση και θα με διευκολύνουν να αναφέρω τη σοβαρότητα του προβλήματος. Νομίζω ότι τα στοιχεία το καταδεικνύουν. Συμφωνούμε όλοι από αυτού. Επίσης αναφέρθηκε από το ΕΛΚΑ ότι πρέπει να τονίσουμε ότι η συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία συμβάλλει στην οικονομική αποδοτικότητα και ότι μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να αναφερθεί. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι με μια πολύ μικρή επένδυση στην ε, αμοιβή αυτών που ασχολούνται με την ανατροφή και τη φροντίδα μπορούμε να κερδίσουμε πολλά. Επίσης ε, οι οικιακά εργαζόμενες, βεβαίως. Υποτιμάται και είναι αόρατη αυτή η εργασία. Και άλλα βασικά στοιχεία, η εκπαίδευση, για θέματα ισότητας που σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να δρούμε και προληπτικά σε πολλούς κλάδους και τομείς οικονομικής δραστηριότητας βλέπουμε να είναι σχεδόν αποκλειστικά άνδρες. Ενώ σε άλλους που είναι υποτιμημένοι και δεν φαίνονται είναι κυρίως γυναίκες, εργάζονται κυρίως γυναίκες. Βεβαίως, ε, πολλές εργασίες οικιακές, φροντίδας και ανατροφής δεν αμείβονται. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε να ζητήσουμε ένα μισθό, αποδοχές για τις φροντίδες αυτές, να έχουν όλοι δικαίωμα στην παροχή φροντίδας. Αυτό είναι το βασικό. Με βεβαίως συνυπευθυνότητα. Φυσικά. Δεν έχουν δικαιώματα μόνο οι μητέρες αλλά και οι πατέρες και βεβαίως και οι κοινοφελείς ε, υπηρεσίες. Οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν το ρόλο τους και ξέρουμε πόσο εθίγησαν από τις πολιτικές λιτότητας τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως όλα αυτά τα σημειώνω και στις περαιτέρω συνεδριάσεις που θα κάνουμε θα τα κάνουμε ακόμη και συγκεκριμένα και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα τα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτούς που καταγγέλουν ε, κακώς κείμενα των καταγγελτών προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών. Επί της ουσίας είναι αρμόδια η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Να δώσω το λόγο στη Σοφία Ριμπέρου που αντικαθιστά τον κύριο ε, Νταβίτ Κάζα. Τρία λεπτά, Σοφία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά αφού αντικαθιστώ τον David Κάσα. Για τον εισηγητή, λοιπόν, σκοπό του σχεδίου γνωμοδότηση. είναι να ενημερώσει η Επιτροπή μα ε, την ε, Επιτροπή Γιούρη, με πληροφορίε σχετικά με θέματα μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προ το δημόσιο συμφέρον, των αποκαλύπτουν εμπιστευτικέ πληροφορίε επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών. Στο σχέδιο γνωμοδότηση υπογραμμίζουμε πώς βοηθούν ε, οι καταγγέλτες να προληφθούν περιπτώσεις διαφθοράς σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και όχι μόνο στον χώρο εργασία. Ο Ντεβιτ Κάσα πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξουμε την ε, δημόσια εικόνα των καταγγελτών, να υπογραμμίσουμε πόσα ωφέλη έχει μια πρόορη προειδοποίηση στην πρόληψη της ε, διαφθοράς και των καταχρήσεων και πώς βοηθά να ενημερώνεται ο κόσμος για τις δράσεις αυτές. Είναι σημαντικό αυτό στη δημοκρατική λογοδοσία. Μία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι ένα στου τρει πολίτε ισχυρίζεται ότι η μη προστασία των καταγγελτών αποθαρρύνει ανθρώπου από το να καταγγείλουν περιπτώσει απάτη. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μέτρα προστασία εργαζομένων που εντοπίζουν και καταγγέλουν παρατυπίες ε, στο εργασιακό τους περιβάλλον, ε, διότι φοβούνται αντίπεινα, είτε ενεργά είτε παθητικά. Ε, είτε δηλαδή απόλυση είτε μη ε, προαγωγή σε περίπτωση ή αντίπεινα από ε, συναδέλφους. Αυτός ο παράγοντας είναι πολύ σημαντικός διότι αποθαρρύνει πολλούς από το να καταγγέλνουν οτιδήποτε. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η προστασία των καταγγελτών έχει αναγνωριστεί από όλα τα μεγάλα διεθνή εργαλεία αντιμετώπισης της αυθόρας. Υπάρχουν όμως τεράστιες διαφορές ακόμα μεταξύ των κρατών μελών. Ορισμένα εξακολουθούν να μην έχουν καμία νομοθεσία. Η διαφθορά είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον κόσμο σήμερα. Είναι ευρέω δεδομένη παντού. Αυτό έδειξε και το πρόσφατο σκάνδαλο με τα έγγραφα του Παναμά. Επηρεάζει αρνητικά ε, τους πολίτες των εν λόγω χωρών. Επαρεμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμού σε πολλά πεδία και δημιουργεί πρόβλημα στους ε, και αποτελεί και παραβίαση των ε, κανόνων ε, του εργατικού δικαίου. Οδηγεί ορισμένε φορέ σε αβέβαιη απασχόληση και σε κακέ συνθήκες εργασίας. Ο Ντεβίτ Κάσα θέλει να υπενθυμίσει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι οι καταγγέλτε δεν είναι καλοπροαίρετοι, οπότε θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη σε περίπτωση ψευδών ε, καταγγελιών ή καταγγελιών που γίνονται ως αντίπεινα ή ως εκδίκηση. Θα δώσω τώρα στο στιώδη συγητή ε, την, ε, το λόγο στην θέση του Γιώργου Παλάση, κυρία Γιονγκέριος. Και προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 12 η ώρα 26 2017, είπε ο Ο κύριος Μπάλας ζητά συγγνώμη που δεν μπόρεσε να παρευρίσκεται εδώ σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κάσα για την πρότασή του και αυτό συμμερίζεται την άποψή του ότι τι τελευταίε δεκαετίε οι καταγγέλτε έχουν διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο για την αποκάλυψη πληροφοριών που σχετίζεται με σημαντικά σκάνδαλα διαφθορά ή ε, μαζική φοροδιαφυγή. Ε, ή ε, χρηματοοικονομικών οργανισμών παραβιάζουν ε, εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πιστεύει ότι σε αυτή τη γνωμοδότηση της ΣΕΜΠΛ θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη. Ε, για να του πούμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο που θα προσφέρει κάποια προστασία των καταγγελτών στο πλαίσιο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων πολύ ενδιαφερόμενοι, πολλές ΜΚΟ ήδη έχουν ε, προτείνει διάφορα μέτρα και κατευθυντήρες γραμμές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των καταγγελτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν κ. Σπέθα να υπογραμμιστούν κάποιες πτυχές. Πρώτον, όπως ανέφερε ήδη η συγητής, η προστασία από οποιοδήποτε αντίπεινα ή διακριτική μεταχείριση θα πρέπει να διασφαλίσετε στον χώρο εργασίας σε περίπτωση κυρώσεων, για παράδειγμα τιμωριών, μείωση καθηκόντων, η παρενόχληση. Η εμπιστευτικότητα και η ανωνυμία των καταγγελτών τη ταυτότητά του, των δραστηριοτήτων του πρέπει να δεσφαλίζεται. Εφόσον δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι ψευδεί οι πληροφορίε που αποκάλυψαν. Οι κανόνες που διέπουν την προσωπική προστασία των καταγγελτών και των οικογενειών τους πρέπει επίσης να εφαρμόζονται σε περίπτωση κινδύνου της ζωής τους. Τέλος, ο κύριος ε, Μπαράς θα ήθελε να υπογραμμίσει ε, τους μηχανισμούς ε, αναφοράς που θα πρέπει να υπάρχουν εντό του χώρου εργασία, αλλά και εντό των ρυθμιστικών αρχών όπου η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών αν αυτή δεν είναι δυνατή θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ε, αυτόνομος ευρωπαϊκός οργανισμός που θα διερευνά την ποιότητα των πληροφοριών που έχουν δοθεί από τους καταγγέλτες. Ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής λοιπόν θα μπορούσε επίσης να αναλάβει μια επιπλέον ευθύνη για το θέμα αυτό και πόρους ώστε να ε, βοηθά ε, ειδικευμένους οργανισμούς για αποκαλύψη τέτοιων πληροφοριών δεν έχουμε ανθρώπους από το ΙΣΕΡΙ ε, ε, το οπότε δίνουμε στην κυρία Μπόλμαν από την ΚΟΕ. Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το σημαντικό θέμα. Ε, πιστεύω πως Αυτές οι καταγγελίες είναι ο πιο, ένας από τους πιο αποτελεσματικούς, αν όχι αποτελεσματικότερος τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς αυτές τις ε, παρατυπίες. Υπάρχουν περιπτώσεις ε, υπαλλήλων που κατήγγυλαν παρατυπίες είτε στους ε, ανωτέρους τους είτε στα μέσα ενημέρωσης. Το 2016 υπήρχαν 2.400 καταγγελίες σε 114 χώρες. Στην Ιρλανδία υπάρχουν τρεις, ε, από όσο ξέρω, ε, έρευνες που διεξάγονται αυτήν την ε, περίοδο που βασίζονται σε καταγγελίες τέτοιου τύπου. Πολλές φορές οι κατηγορίες αυτές αφορούν κακοποίηση ανηλίκων από την αστυνομία, από τον χώρο της πολιτικής. Και σε μία από αυτές τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι μία από αυτές τις καταγγελίες ήταν ε, ψευδής και σκοπό είχε να καταστρέψει τη φήμη του ε, προσώπου. Στην έκθεση χρειάζεται να συμπεριληφθεί μία εγγύηση για την ασφάλεια εκείνων που δείχνουν το θάρρος να καταγγείλουν αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες και τις ε, παραβιάσεις οι καταγγέλτες αυτοί είναι απαραίτητοι, διότι προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον, αυξάνουν την ακαιρεότητα και την λογοδοσία τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτοί οι καταγγέλτες παίρνουν ε, μεγάλο ρίσκο κάνοντας αυτές τις καταγγελίες. Το κόστος είναι προσωπικό, επαγγελματικό, γενικότερο. Χρειάζεται λοιπόν να δείξουμε όλοι μας τη στήριξη σε αυτούς ε, τους ανθρώπους. Αυτό έχει αναγνωριστεί και από διεθνεί οργανισμού η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στις περισσότερες από αυτές ε, τις ε, συμβάσεις και πέρυσι τα Ηνωμένα Έθνη πρότειναν ενισχυμένη προστασία για τους καταγγέλτες ε, με την αντίστοιχη έκθεση. Από όσο γνωρίζω τα κράτη-μέλη δεν έχουν δείξει επαρκή προθυμία για να προστατεύσουν τους καταγγελτές. Έξι μάλιστα από, τις, από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει καμία προστασία εδώ πρέπει να λάβουμε υπέψη μεν και την επικουρικότητα, αλλά να κοιτάξουμε τις ε, καλύτερες πρακτικές τόσο στην Ένωση όσο και παγκόσμια και να προωθήσουμε την καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος εργασίας όπου οι υπάλληλοι θα αισθάνονται άνετα ε, και θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τα παράπονά τους ή τις ανησυχίες τους εάν αυτά προκύψουν. Πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα όπου οι πολίτες θα ε, τολμούν να καταγγέλουν τα κακό κείμενα. Και είναι πολύ σημαντικό επίση, ε, μπορείτε να συντομεύετε, λέει ο Πρόεδρο. Είναι λοιπόν εξίσου σημαντικό να προστατεύονται οι καταγγέλτε ε, και από την κοινωνία και από τα μέσα ενημέρωση. Πρέπει να αλλάξει λοιπόν η νοοτροπία, η κουλτούρα και όχι μόνο η νομοθεσία. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Τέρι Ράιν και για του πράσινου. Για δύο λεπτά αν μπορείτε. Θα προσπαθήσω, θα κάνω ό,τι μπορώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο και καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Κάσα. Ίσως η κυρία Ριμπέιρο μπορεί να του μεταφέρει τις ευχαριστίες μου. Είναι πολύ καλό σχέδιο έκθεση, είναι μια πολύ καλή αφετηρία και συζήτηση, πιστεύω. διότι οι καταγγέλτες έχουν έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για τις ε, περιπτώσεις ε, καταγγελτών που αποκάλυψαν ε, θέματα που αφορούν την παγκόσμια κοινότητα, αποκάλυψαν απάτες, ε, όμως επίσης σας μην ξεχνάμε και τους καταγγέλτες που ε, κατήγγυλαν παράνομες δραστηριότητες, εγκληματικές δραστηριότητες, ε, επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για τη δική μας ομάδα των Πρασίνων, καταρχάς τα μέτρα προστασίας να συμπεριλαμβάνουν και το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, να είναι υποχρεωτικά για τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν, υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Επίσης, ε, πρέπει να αναφερθούν οι κλιματικές δραστηριότητες, αλλά και οι παρατυπίες στον ε, χώρο εργασίας, αντιδιαλοντογική συμπεριφορά. Και για μας είναι επίσης πολύ σημαντικό να προστατεύονται οι καταγγέλτες και οι οικογένειές τους και να συμπεριλαμβάνονται κυρώσεις για πιθανή ε, παρενόχληση και εκφοβισμό μετά από μια καταγγελία. Τέλος, χρειάζεται να κληθούν τα κρατημέλη να δημιουργήσουν νομοθεσία για την προστασία των καταγγελτών, όμως και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα παρικούς προστασία στους καταγγέλτες. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Ε, συζητήσαμε πέρυσι σε αυτήν την Επιτροπή της καταγγελίας για την αφήλωτη εργασία. Οπότε θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε εδώ και κάποια άρθρα για τους καταγγέλτε ό,τι θέμα αφορά αυτήν την Επιτροπή, νομίζω πως πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τη διάσκεταση της προστασίας των καταγγελτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Μαχτάν για το ΙΕΝΕΦ. Ε, για μια φορά ε, θα σας βοηθήσω να καλύψω την καθυστέρηση. Ε, για το θέμα αυτό η ομάδα μου δεν έχει άποψη. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα με βοηθήσει να καλύψω όλη την καθυστέρηση. Αλλά εν πάση Να ξαναδώσω το λόγο και πάλι στην κυρία Ριμπέιρο. Α, δεν έχει τίποτα να προσθέσει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Αλλά για το επόμενο θέμα ο εισηγητή μα δεν είναι εδώ. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή 5 λεπτών. Ελπίζω όχι περισσότερο. Γιατί ο εισηγητή ε, ξέρει ότι το θέμα του είναι για τι 11 Πέντε λεπτά, σας παρακαλώ μην φύγετε, για να μπορέσουμε να ξαναρχίσουμε μόλις ε, τη συνεδρίασή μας μόλις ε, εμφανιστεί ο εισηγητής.

Okay, Σας προτείνω να συνεχίσουμε. Ε, ε, έχουμε ένα προβληματάκι απουσία του εισηγητή, διότι είχε ένα πρόβλημα με την πίστη του, οπότε πιθανώς να μην έρθει. Οπότε προτείνω να αλλάξουμε λίγο τις εργασίες μας από ό,τι είχε προγραμματιστεί. Θα ξεκινήσουμε ακούγοντας πρώτα απ' όλα την Κομισιόν, λοιπόν, και μετά θα περάσουμε στη συζήτηση. Για αυτό το θέμα λοιπόν που αφορά το κοινό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές ε, σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο. Βάσει διαφόρων δειγμάτων ε, δίνω το λόγο στην Κομισιόν. Σας ευχαριστώ που δείξατε τόση ευελιξία σε σχέση με το ότι είχε προγραμματιστεί στην αρχή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Σε ό,τι αφορά την πρότασή μας για τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά με βάση στοιχεία, θα ήθελα να πω καταρχάς δύο λόγια για το πλαίσιο του κανονισμού αυτού. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι αξιόπιστες και ε, επίκαιρες στατιστικές είναι πάρα πολύ σημαντικές για την χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής. Αφορούν άμεσα και το ευρωπαϊκό εξάμεινο, αλλά και όχι μόνο, διάφορους τομείς πολιτικής και αντιμετωπίζουν επίσης την ανάγκη έβρεσης ερευνητών και γενικότερα χρηστών αυτών των πληροφοριών. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται σε πολιτικές που αφορούν την κοινωνία και τις εξελίξεις ε, σχετικά με αυτή στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες. Θέματα όπως η ανάπτυξη, οι θέση απασχόλησης, η πρόσβαση στην απασχόληση, η φτώχεια και ο αποκλεισμός, αποκλεισμό, οι ανισότητες και η άνεση κατανομή δεξιοτήτων, η κοινωνική προστασία, η ισότητα των φύλων, ε, οι ορισμένες κοινωνικές ομάδες, όλα αυτά μπορούν να περιγραφούν με αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και επίκαιρα στατιστικά στοιχεία. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να παρέχονται πληροφορίες για έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις ε, ε, προτεραιότητες που αλλάζουν συνεχώς να προσαρμόζονται και στους δημοσιονομικούς διαθεσιμούς πόρους. Για να ανταπεξέλθουμε λοιπόν σε αυτήν την ανάγκη για αξιόπιστα και ε, επίκαιρα στατιστικά στοιχεία, συνεργαζόμαστε με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των κρατών μελών εδώ και πολλά χρόνια, έτσι ώστε να εξυγχρονίσουμε τα κοινωνικά στατιστικά στοιχεία. Ο κανονισμός πλαίσιο λοιπόν που έχετε ενώπιόν σας είναι το αποτέλεσμα αυτής της κοινή προσπάθειας με τα κράτη-μέλη και με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτός ο κανονισμός, εφόσον εγκριθεί, θα γίνει ένα εργαλείο με το οποίο θα εξυγχρονιστεί η στατιστική επιστήμη. Θα έχουμε καλύτερα στατιστικά στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν με τη σειρά τους να χαράξουμε καλύτερη πολιτική. Αυτό που κάνει ο κανονισμός αυτός είναι ότι απλουστεύει την συλλογή δεδομένων, επτά ομάδων δεδομένων. Και το σκεπτικό είναι να τυποποιηθεί τόσο η μεθοδολογία όσο και τα μέσα συλλογής αυτών των δεδομένων. για να μπορούμε να είμαστε ενήμεροι για τις νέες τάσεις και εξελίξεις. Για παράδειγμα, όταν γίνεται λόγος για νέες δεξιότητες στην αγορά εργασίας, χρειαζόμαστε όχι μόνο στατιστικά στοιχεία από έρευνες ε, για το χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και στατιστικά στοιχεία από έρευνε που αφορούν το χώρο εργασίας, την αγορά εργασίας. Υπάρχει λοιπόν ε, μεγάλη γκάμα θεμάτων που αφορούν αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Και φυσικά έχουμε απόλυτη επίγνωση του κόστους και του διοικητικού φόρτου που θα προκύψει από αυτές τις πρόσθετες ανάγκες. Γι' αυτό στον κανονισμό αυτό προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό χρησιμοποιώντας σύγχρονους τρόπους συλλογής δεδομένων, σύγχρονες μεθόδους, σύγχρονα εργαλεία, προωθώντας την χρήση του μεγάλου όγκου δεδομένων, των διοικητικών δεδομένων, διαφόρων τύπων δεδομένων Προσπαθήσαμε επίσης να δώσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στο κόστος, δηλαδή να τυποποιήσουμε τις προθεσμίες υποβολής δεδομένων, ε, την, το χρόνο συλλογής των δεδομένων κτλ. Και τέλος υπάρχουν ορισμένες ε, οικονομικές διατάξεις έτσι ώστε οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες να έχουν οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να υλοποιήσουν όλες τις διατάξεις του κανονισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους στόχους του κανονισμού πλαισίου, θέλουμε να βελτιωθούν τα χρονοδιαγράμματα. Οι προθεσμίες δηλαδή που οι προθεσμίες υποβολής των ε, στατιστικών στοιχείων ε, να συνδεθούν με, την, ε, με τις προθεσμίες πολιτικής. Για παράδειγμα, να συνδεθούν με τις προθεσμίες του Ευρωπαϊκού Ξαμήνου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλα προβλήματα στο συγχρονισμό των χρονοδιαγραμμάτων πολλές φορές στατιστικά στοιχεία συλλέγονται δύο χρόνια πριν από τη στιγμή που αναλύονται. Γι' αυτό λοιπόν ο κανονισμός ε, αυτός αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Μετά, ε, συγκρισιμότητα στοιχείων, συλλογή των στοιχείων, χρόνο συλλογής, είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά έτσι ώστε οι πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο να είναι αποτελεσματικές και να υπάρχει η μεταχείριση των κρατών μελών. Είναι πάρα πολύ σημαντική επίσης και η ευελιξία. Είναι και στόχος του κανονισμού. Όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε αυξημένα αιτήματα για παροχή δεδομένων και έχουν αλλάξει προτεραιότητες. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε ευελιξία και να δείξουμε ότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Η ευελιξία τι σημαίνει. Σημαίνει καταρχάς ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να μετρήσουμε τις νέες τάσεις, τα νέα φαινόμενα. Και αυτά τα φαινόμενα είναι ε, διάφορα. Για παράδειγμα, υπάρχουν, πια, πού είναι τα όρια ανάμεσα στην απασχόληση και στην αυτοαπασχόληση. Ε, ποιος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ε, αληθινός ε, και ποιος έχει μεν αυτή την ιδιότητα, αλλά έχει έναν μεγάλο πελάτη από τον οποίο εξαρτάται οικονομικά. Μετά πρέπει να δίνουμε πληροφορίες για τις νέες τάσεις στην εργασία, δηλαδή συμβόλαια, συμβάσεις μηδενικών όρων εργασίας ή ελάχιστων όρων εργασίας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε τις κατάλληλες στατιστικές για να μπορούμε να αναλύσουμε αυτές τις τάσεις. Και παρομοίως για την ανάγκη ε, που υπάρχει να δώσουμε βάση στους ε, ηλικιωμένους, να ε, φροντίσουμε να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Τώρα και σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα της υγείας των ηλικιωμένων, χρειάζεται και εδώ να έχουμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία αλλά όχι μόνο για τους ηλικιωμένους και για άλλες ομάδες του πληθυσμού. Για παράδειγμα τα άτομα με αναπηρία, τους μετανάστες. Ε, θέματα ένταξης επίσης. Ένταξης ε, μεταξύ άλλων και στην αγορά εργασίας. Είναι πολύ σημαντικά και πολύ επίκαιρα τελευταία, ιδιαίτερα εν ώψη των δεδομένων των εξελίξεων. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργήσουμε μια τελείως ε, καινούρια στατιστική βάση που θα μας επιτρέπει να μετρήσουμε αυτά τα φαινόμενα και να ακολουθούμε ε, τις εξελίξεις ε, με την πάροδο του χρόνου. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κωδικοποιήσουμε αυτήν την ε, βάση δεδομένων στις ήδη υπάρχουσες βάσεις. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχουν ε, οι κατάλληλες δομές έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να ε, μετρήσουμε αυτά τα νέα φαινόμενα. Τώρα, ε, ας μιλήσουμε για αυτές τις μεταβλητές. Στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας του Συμβουλίου έχουν γίνει έντονα συζητήσεις γι' αυτό. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα σε αυτόν τον κανονισμό. Το πρώτο είναι η αγορά εργασίας, οι συνθήκες διαβίωσης για παράδειγμα. Μετά, υπάρχουν κάποια πολύ βασικά ζητήματα σε κάθε τομέα, για παράδειγμα, συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Συνθήκες ε, διαβίωσης, στέγαση φτώχεια, ανέχεια. Αυτά ε, αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης. Έχουμε προβλέψει και ένα τρίτο επίπεδο στο παράρτημα 1 του κανονισμού αναφέρεται αυτό με λεπτομέρειες, αν θέλετε να το διαβάσετε. Εκεί καλούμε τους νομοθέτες να εντοπίσουν τα συγκεκριμένα θέματα που ε, χρήζουν αλλαγή πολιτικής. Θεωρούμε πως αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Γι' αυτό και έχουμε καλέσει τον νομοθέτη να διορθώσει το σημείο αυτό στο κανονισμό και να το πλησιώσει έτσι ώστε να καθορίζονται σαφώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούμε να αναπτύξουμε αυτές τις πολιτικές. Πρέπει λοιπόν πρώτα να διορθώσουμε τον κανονισμό και γι' αυτό έχουμε προβλέψει πράξεις κατά εξουσιοδότηση για να εξελιχθεί έτσι το θέμα και έχουν προβλεφθεί επίσης δράσεις για να μειωθεί το κόστος και ε, ο φόρτος που θα συνοδεύει αυτή την εξέλιξη. Χρειάζεται αυτή η εξέλιξη. Είναι αναγκαία γιατί μόνο έτσι μπορούν να υλοποιηθούν ε, οι νέες προτάσεις. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Και τώρα ασταθούμε και στις μεταβλητές και το ρόλο τους. Οι μεταβλητές έχουν ως εξή Εφόσον προσδιοριστεί ένα συγκεκριμένο θέμα, καθορίζουμε ουσιαστικά οι εμπειρογνώμες δηλαδή συζητούν και καθορίζουν τις μεταβλητές που είναι αντιπροσωπευτικές ώστε να δοθεί η μέτρηση για το θέμα αυτό που ζητούν οι υπευθύνοι χαράξεις πολιτικής και οι νομοθέτες. Οι μεταβλητές ε, χαρακτηρίζονται από το εξής. δύο μεταβλητές μπορεί να φαίνονται ε, ίσες αριθμητικά ένα και ένα ας πούμε να είναι αλλά η μία μπορεί να σημαίνει ένα να αντιστοιχεί σε ένα, δύο ή δέκα ερωτήματα οπότε συνεπώς δύο μεταβλητές δεν είναι απαραίτητα ίδιες όσον αφορά τις συνέπειες τους και φυσικά και ο αριθμός των ερωτημάτων έχει συνέπειες και αποτελέσματα όσον αφορά τη διάρκεια της συνέντευξης και το τι ζητείτε να απαντήσει κάποιος. Επίσης υπάρχουν διαφορές στις συχνότητες. Ορισμένες μεταβλητές ε, θα έχουν τριμηνία συχνότητα, άλλες ετήσια συχνότητα, άλλες οκταετή συχνότητα. Οπότε και εδώ υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μεταβλητών αυτών. Και τέλος, Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ αυτού που ονομάζουμε τεχνικές μεταβλητές και λοιπές μεταβλητές. Οι τεχνικές μεταβλητές είναι αυτές για τις οποίες δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε τον ε, ρωτηθέντα. Για παράδειγμα την ημερομηνία της συνέντευξης, τον τύπο της συνέντευξης, ε, κατά πόσο είναι πρόσωπο με πρόσωπο, ε, η υπολογιστή, η διαδικτύου. Όλα αυτά είναι μεταβλητές, ε, αλλά δεν τις ε, συλλέγουμε εμείς. Τι σημαίνει αυτό. Ότι στον κανονισμό δεν υπάρχει λόγος να οριστεί ο αριθμός μεταβλητών, ούτε να περιοριστεί ο αριθμός μεταβλητών κατά οποιονδήποτε τρόπο. Θεωρούμε εμείς ότι οι εμπειρογνώμονες είναι εκείνοι που θα πρέπει να το συζητήσουν και να καταλήξουν στις πιο αντιπροσωπευτικές μεταβλητές. Το να καθορίσουμε αυστηρά ένα συγκεκριμένο αριθμό μεταβλητών ε, αντίκειται στο βασικό ρόλο της νομοθεσίας αυτής, δηλαδή του να μπορέσει ουσιαστικά να ανοιχνεύσει νέα φαινόμενα με τρόπο ευέλικτο, όπως το ανέφερα νωρίτερα. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική σκέψη ε, όταν μιλάμε για θέματα ευελιξίας. Από αυτό προκύπτει ότι εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει ένα σωστό θέμα ανάλυσης όπου εμείς λέμε ε, για ποιο θέμα θέλουμε πληροφορίες και πώς θέλουμε να το πλαισιώσουμε. Αυτό το λέμε εμείς στους νομοθέτες. Γι' αυτό έχουμε συμπεριλάβει αυτά τα αναλυτικά ζητήματα σε αυτό το σχέδιο κανονισμού. Λοιπόν, τώρα... Ε, πριν μπω στις κύριες ε, τροπολογίες που έχουν γίνει, να πω δύο λόγια για ορισμένα ζητήματα τα οποία συζητάμε στην ε, ομάδα εργασίας στο Συμβούλιο σχετικά με τις στατιστικές. Ανέφερα τον αριθμό των στόχων αυτού του, αυτής της νομοθεσίας. Πρώτα απ' όλα, ε, η κατάλληλη χρονική στιγμή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν θέλει κανείς να συνδέσει τα στατιστικά στοιχεία με διάφορα άλλα πλαίσια όπως το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που μας ζητά να τρίσουμε για παράδειγμα την κοινωνική επίπτωση ε, κάποιων πολιτικών. Εκεί λοιπόν πρέπει να βελτιώσουμε το χρονοδιάγραμμα, το χρονοδιάγραμμα και το πόσο επίκαιρα είναι τα στοιχεία. Ανέφερα αυτό για τα εισοδήματα και εδώ πολλά κράτη-μέλη ισχυρίζονται ότι ε, είναι πολύ δύσκολα τα χρονικά περιθώρια που βάζουμε ως έγκαιρα ε, σε αυτή τη νομοθεσία. Στην έρευνά μας για τις ε, συνθήκες διαβίωσης προτείνουμε τα στοιχεία για το έτος αναφοράς νη που συλλέγονται στο έτος νη συν 1 να είναι διαθέσιμα στο τέλος του νη συν 1 ώστε να ε, με το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Εξάμενου. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε πολλά κράτη-μέλη. Το δεύτερο ζήτημα είναι η ευελιξία. Όπως ε, είπα, βρίσκεται στο επίκεντρο του κανονισμού αυτού. Για να μετρήσουμε, να αξιολογήσουμε τα νέα φαινόμενα, και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε γρήγορα στα νέα αιτήματα των νομοθετών και των υπευθύνων χαράξη πολιτική, ε, αυτή η ευελιξία είναι απαραίτητη. Σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την έκταση της ευελιξίας αυτής. Ειδικότερα, όπως εξήγησα προηγουμένως, πιστεύουμε ότι το σωστό επίπεδο είναι λεπτομερή θέματα και όχι μεταβλητές σε αυτή την νομοθεσία. Και δεν θα πρέπει να ορίσουμε αυστηρά ένα συγκεκριμένο αριθμό μεταβλητών που θα συζητούν οι εμπειρογνώμονες, λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα την αντιπροσωπευτικότητα. Ένα τρίτο ζήτημα σχετίζεται με το πώς συμπεριλαμβάνονται οι διάφορες έρευνες για τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά σε αυτό τον κανονισμό. Τι έχουμε κάνει εμείς, έχουμε φροντίσει να προβλέψουμε, να καλύπτονται αυτές οι δύο έρευνες από αυτόν τον κανονισμό, δίνοντας επαρκή χρόνο στους υπευθύνου ε, στατιστικής ε, να συνεργαστούν και να εξυγχρονίσουν αυτές τις ε, δύο έρευνες, βασίζοντάς πάνω σε νέα στοιχεία, διοικητικά στοιχεία, μεγάλα στοιχεία, νέα εργαλεία, μοντέλα ώστε να μειωθεί σημαντικά το κόστος των ερευνών αυτών. Ε, προβλέπεται δεκαετής περίοδος για την υλοποίηση αυτού του κανονισμού για έρευνες ε, για τα νοικοκυριά. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να είμαστε τόσο φιλόδοξοι ώστε να γίνει το έργο αυτό εξυγχρονισμού. Ένα τέταρτο ζήτημα τι γίνεται με το πάνελ ε, για την έρευνα των συνθήκων διαβίωση. Οι χρήστε ζητούν ε, το χρονοδιάγραμμα αυτό να επεκταθεί από τα 4 στα 6 χρόνια για την έρευνα αυτή των οικοκυριών και τι συνθήκε διαβίωση του, ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις πορείες ε, προσώπων και νοικοκυριών καθώ βγαίνουν από τη φτώχεια. Γιατί ξέρετε, το να βρει κάποιο δουλειά δεν σημαίνει ότι βγήκε από τη φτώχεια. Μετά τίθεται το πέμπτο ζήτημα της συγκρισιμότητας. Γενικότερα, στη συγκρισιμότητα χρησιμοποιούμε την προσέγγιση αποτελεσμάτων. Δηλαδή, ε, θέτουμε τους ίδιους ορισμούς και αφήνουμε τα κράτη-μέλη να τους εφαρμόσουν. ώστε να υπάρχει εγγενή συγκρισιμότητα των δεδομένων. Αυτό λειτουργεί σε κάποιου τομεί, είναι ο γενικό μα κανόνα, αλλά σε κάποιου ε, τομεί και βάσει μελετών, και τώρα αναφέρομαι ειδικότερα στην απασχόληση και την ενεργεία, τα νούμερα δείχνουν ότι η σειρά των ερωτημάτων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά έναν βασικό δίκτυο όπως ε, το δίκτυο ενεργείας. Τέτοιες συζητήσεις κάνουμε αυτή τη στιγμή στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Δεν έχουμε δει τις, ε, έχουμε δει τροπολογίες ε, στην αρχική έκθεση του ε, εισηγητή και αυτές που έχετε υποβάλει εσείς. Θα θέλαμε φυσικά να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή και όλους τους βουλευτές και όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για αυτές τις τροπολογίες. τις ερμηνεύουμε ως ισχυρή υποστήριξη των στόχων που ανέφερα νωρίτερα. Ειδικότερα της ευελιξίας, του έγκυρου χαρακτήρα και της συγκρισιμότητας. Τώρα. Είδαμε τώρα μερικές συγκεκριμένες τροπολογίες θα μπορούσα να σας πω ποια είναι η γνώμη μας για αυτές, εκτός αν ε, προτιμάτε πρώτα να γίνει συζήτηση και μετά να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας που ήταν ιδιαίτερα αναλυτική. Αν έχουμε χρόνο μετά τις παρεμβάσεις θα σας ξαναδώσουμε το λόγο. Καταρχάς Μόλις έλαβα ένα μήνο από τον εισηγητή μας, ο οποίος ε, μας ζητάει συγγνώμη για την απουσία του, για λόγους ε, ανεξαρτήτους ε, της θελήσεώς του. Έγιναν λοιπόν δύο συνεδριάσεις των σκιωδών και τονίζει ότι οι συζητήσεις υπήρξαν επικοδομητικές και διαφάνηκαν σαφώς οι δυνατότητες συμβιβασμών ευχαριστεί τους Κιώδης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βοήθεια που του έχουν δώσει για μια σειρά από θέματα, κυρίως για τεχνικής φύσης ζητήματα. Λοιπόν, δεν βλέπω κανένα για το ΕΛΚΑ. Να δώσω το λόγο στην Αγνιές Γιόγκερης για, το, για τους σοσιαλιστές. Ωραία. Τώρα από πλευρά του κυρίου Πυρίνσκι, που και εκείνος απουσιάζει, Ευχαριστώ λοιπόν εκ μέρους του την, ε, τον εισηγητή για την επικοδομητική του προσέγγιση. Θα τον ευχαριστούσα αν ήταν παρόν και ο εισηγητής. Να αναφερθώ τώρα στις τροπολογίες που υπέβαλαν συνάδελφοι της ομάδας μου. Διευκρινίζουν τους κύριους στόχους μας. Θέλουμε την μεταρρύθμιση των ε, κοινωνικών στατιστικών, όπως προτείνεται από το, τον κανονισμό πλαίσιο, αλλά θέλουμε να βοηθήσουν την βελτίωση του καθορισμού των πολιτικών στόχων και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τομέα αυτό. Θέλουμε λοιπόν καλύτερα στοιχεία για να μας στηρίζουν. Δεύτερον πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει σαφήνεια για τη συμβατότητα του νέου κανονισμού πλαισίου με τον υπάρχοντα κανονισμό που θα συνεχίσει να ισχύει για ε, συλλογή στοιχείων που δεν θα καλύπτεται σε τομείς που δεν καλύπτει ο νέος κανονισμός. Και θέλουμε να υπάρξουν οι ε, ορισμοί που θέλουμε, που είναι σημαντικοί για τον κανονισμό, για παράδειγμα ποιος είναι ο ορισμός του νοικοκυριού. Επίσης θέλουμε ο τίτλος ενός συγκεκριμένου πεδίου ε, εργατικό δυναμικό να ε, συνδυάζεται με τα στοιχεία για την αγορά εργασίας η, η έρευνα για την αγορά εργασίας λοιπόν συμπεριλαμβάνει πολύ ευρύτερε έρευνε και για επιχειρήσεις. Η πρόταση όπως είναι τώρα, για τον κανονισμό πλαίσιο όμω, αναφέρεται μόνο σε άτομα ή σε νοικοκυριά. Δεν καλύπτει τις έρευνες ε, για τις επιχειρήσεις, όπως λέει η αιτιολογική σκέψη 11. Ο όρος λοιπόν ε, εργατικό δυναμικό πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη γνώμη μας με τον όρο αγορά εργασίας. Έχουμε τροπολογίες για να διευκρινίσουμε το άρθρο 3, τα κοινά αναλυτικά θέματα και τα θέματα που αφορούν όλες τις, όλους τους τομείς. Αυτό θα διευκρινίσει την κατάσταση στο παράρτημα 1. Και τέλος, ότι Θέλουμε να είναι βαθιά αυτή η μεταρρύθμιση, αλλά αυτό θα έχει ένα κόστος. Καλούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότηση προς τα κράτη-μέλη, όπου χρειάζεται για να εφαρμοστεί αυτός ο νέος κανονισμός. Και τέλος, η ομάδα μου στηρίζει τις τροπολογίες του εισηγητή που ε, αναφέρονται στην ανάγκη για κατεξοδότηση πράξη και όχι εφαρμοστικέ πράξει. Γιατί έτσι το Κοινοβούλιο θα μπορεί να ελέγξει καλύτερα την εφαρμογή του κανονισμού πλαισίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ίσια, η κυρία Τρεμπέσιου. Ευχαριστώ. Και στην προηγούμενη συζήτηση για το θέμα αυτό στην Επιτροπή είπα ότι εγώ και η ομάδα μου υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό την πρόταση της Κομισιόν. Έχω μικρή εμβέλεια ε, ε, παρατηρήσεις που αφορούν το κόστος των μελετών και την εμπιστευτικότητα των στοιχείων. Η ομάδα μου, όπως σας είπα λοιπόν, είναι ικανοποιημένη από το κείμενο αυτό. Θέλουμε να υπάρχουν σαφή στοιχεία και συγκρίσιμα για όλες τις χώρες που να βοηθήσουν και τους επιστήμονες ε, και τους οικονομικούς παράγοντες και τους πολιτικούς για να εξάγουν τα σωστά συμπεράσματα. Υπάρχουν ορισμένε τροπολογίε που είναι περισσότερο πολιτικοποιημένε. Ε, δεν προσπαθούν να προωθήσουν την ουδετερότητα των στατιστικών, αλλά θέλουν να προωθήσουν πολιτικού στόχου. Ε, για παράδειγμα, ισότητα ή πολιτική για την ισότητα των φύλων. Ε, εδώ δεν είναι η σωστή ευκαιρία για να προωθήσουμε αυτούς τους στόχου Εδώ πρόκειται για πρωτογενή στοιχεία, τα οποία συλλέγονται για να κάνουμε ε, μετά αξιολογήσει. Δεν πρέπει λοιπόν να πολιτικοποιήσουμε το θέμα αυτό. Βεβαίω θα υποστηρίξω λοιπόν την έκθεση, εάν δεν αποκλίνει πολύ από την ε, πρόταση τη Επιτροπή. Δεν θα υποστηρίξουμε προτάσει με τι οποίε δεν θεωρούμε σοβαρέ. Και ελπίζω ότι με τις δικές μας προτάσεις θα επανέλθουμε στην πολύ καλή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Άντε. Ενρίκε Καλβέτ Τσαμπόν. Ευχαριστώ. Η Άλντε υπέβαλε πολλές τροπολογίες. Τώρα δεν θα μπω σε όλες αυτές, αλλά απόλυτα επικοδομητικές. Μας αρέσει ιδιαίτερα αυτό που προτείνει η Κομισιόν. Και επίσης, συμμεριζόμεθα και πολλές από τις προτάσεις βελτίωσης ε, του εισηγητή, στο πνεύμα τους. Τώρα στις ε, διατυπώσεις ε, αποκλίνουμε και να δούμε αν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε σημεία συμφωνίας. Η αφετηρία μας είναι προφανής. Είναι η φράση του Ισραήλ ότι υπάρχουν ψέματα, άθλια ψέματα και στατιστικές. Οι στατιστικές πάντα θα είναι πολιτικό εργαλείο. Ε, δεν γίνεται να μην είναι. Η στατιστική μας επιτρέπει να κάνουμε πολιτική. Έχει πολλές πλευρές που έχουν ε, πολιτική σημασία. Για παράδειγμα, τι ακριβώς θα μετρήσουμε. Τι αποφασίζουμε, να μετρήσουμε το α και όχι το β. Αυτή είναι μια απόφαση πολιτική. Κάτι που επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι οι ορισμοί του τι ακριβώς θα μετρήσουμε. Για μας η στατιστική πρέπει να προωθήσει μια καλύτερη κοινωνία, περισσότερη ισότητα. Αυτό είναι θεμελιώδες. Θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε την Επιτροπή να βελτιώσει την πρότασή τη ε, σε ορισμένα σημεία, αλλά πάντα λαμβάνουμε υπόψη και το κόστος που μπορεί να προκύψει. Και βεβαίως ε, βασιζόμεθα και στην ε, αρχή του ότι το καλύτερο είναι εχθρό του καλού. Άρα δεν πρέπει να έχουμε υπέρμετρε φιλοδοξίε. Η στατιστική είναι επίσης διεθνέ μέσο. Πρέπει λοιπόν αυτά που θα αποφασίσουμε να είναι συμβατό και συγκρίσιμο με τις στατιστικές των διεθνών οργανισμών του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ και άλλων διεθνών οργανισμών. Δεν πρέπει τώρα εμείς να δημιουργήσουμε δικούς μας ορισμούς και να συλλέγουμε πολύ λεπτομερή στοιχεία. Κάτι που πρέπει να περιέχει, να περιέχει κατά τη γνώμη μας το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα είναι ότι πρέπει να βασίζεται με εναρμονισμένες βάσεις και στατιστικές προδιαγραφές. Προφανές και πρέπει οπωσδήποτε να συμμορφούνται με τον κώδικα ε, δεοντολογίας για τις στατιστικές, να συμμορφώνονται λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί και ε, στον τομέα αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Να δούμε πώς συλλέγουν στατιστικά στοιχεία ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ στην Ευρώπη έχουμε απλώς έναν μηχανισμό ο οποίος δεν συλλέγει στοιχεία, ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό, απλώς λαμβάνει τα στοιχεία που συλλέγει ε, ένας τεράστιος αριθμός ε, εθνικών ε, στατιστικών υπηρεσιών. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τις χώρες που δεν έχουν πολύ ανεπτυγμένο στατιστικό σύστημα. Στατιστικούς φορείς δηλαδή, φορείς στατιστικής. Θέλουμε φυσικά το επίπεδο ΝΑΤΣ 2 για τα στατιστικά μας στοιχεία, όπως λέει και η Επιτροπή. Και επίσης, επιτέλους, πρέπει να ορίσουμε επακριβώς τι σημαίνει νοικοκυριό, ποιο είναι ο στατιστικό ορισμό του. Και δεν το κάνουμε, δεν θα κάνουμε και σωστή πολιτική, γιατί θα υπάρχουν διάφορε ερμηνείε και τα στοιχεία που θα συλλέγουμε δεν θα μα βοηθούν. Δεν θέλουμε να υπάρχουν επικαλύψεις με τις στατιστικές ε, της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζα, Έχει ένα ενοποιημένο στατιστικό σύστημα που μπορεί να μα μάθει πολλά. Δεν θέλουμε επικαλύψεις λοιπόν με την ΕΚΤΑΦ όταν συλλέγουμε στοιχεία για την κατανάλωση, γιατί ήδη τα συλλέγει εκείνη. Λοιπόν, τώρα για τις εξαιρέσεις ή για το χρόνο που χρειάζονται τα κράτη-μέλη, δηλαδή για να προσαρμοστούν εξαιρέσεις που πρέπει να χορηγήσουμε στα κράτη-μέλη και πόσο θα, πόσο θα είναι αυτός ο χρόνος, πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά πώς είναι η κατάσταση σε κάθε χώρα. Είναι πολύ τεχνικό το θέμα λοιπόν. Δεν θέλουμε να τους πιέσουμε δεν πρέπει να τους πούμε ότι θέλουμε οπωσδήποτε τώρα να το επιτύχετε. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν ε, ρεαλιστικό. Και βεβαίως θα επιμείνουμε. Εάν γίνουν αλλαγές, μετά από κάθε αλλαγή, δεν θέλω να πω ότι υπάρχει κακή πρόθεση, αλλά υπάρχουν πολιτικές επιπτώσεις. Θεωρούμε ότι φυσικά πρέπει να είναι κατεξοδότηση οι για να μπορεί το Κοινοβούλιο να τις μελετά, και να μπορεί να κατανοήσει εάν χρειάζονται όντως αλλαγές. Δεν πρέπει να το αφήσουμε στα χέρια μόνο των εμπειρογνωμόνων ε, παρά τις ε, ιεσδήποτε καλές τους προθέσεις. Πρέπει να υπάρχει και ένα πολιτικό επίπεδο που να αποφασίζει για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ Γκούε. Η κυρία Λίν Μπόιλαν. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σύγχανα τον εισηγητή παρά την απουσία του για το σχέδιο έκθεσης και τις συμβαστικές τροπολογίες. Νομίζω πως χειρίζεται το θέμα αυτό με τη λεπτότητα και διακριτικότητα που το αρμόζει. Ε, στηρίζω όλες τις συμβαστικές ε, τροπολογίες που λάβαμε μέχρι τώρα και χαίρομαι πάρα πολύ και τον ευχαριστώ και όλες που συμπεριέλαβα τις δικές μας προτάσεις. Νομίζω ότι για να αντιμετωπίσουμε με πτυχία τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται τα κατάλληλα στατιστικά στοιχεία έτσι ώστε να μετρήσουμε ε, με ακρίβεια το τι συμβαίνει. Γι' αυτό χρειάζεται όμως προσοχή στην αρχή της επικουρικότητας και σε γενικές γραμμές ε, συμφωνώ με την ε, πρόταση αυτή. Χρειάζεται ένα ευρύτερο πλαίσιο για τις στατιστικές υπηρεσίες. Έχω όμως κάποιες επιφυλάξεις για ορισμένε πτυχές του κανονισμού. Δηλαδή, δεν είμαι υπέρ της εναρμόνισης της εισαγωγής στοιχείων για τις ε, έρευνες σχετικά με το εργατικό δυναμικό. Θεωρώ πως εδώ δεν ακολουθείται η αρχή της επικουρικότητας. Επίσης, ε, δεν είμαι μόνη μου, έχουν και άλλα μέλη εκφράσει τις ανησυχίες τους για αυτό το σημείο. Επίσης, ε, οι χώρες της Ευρωζώνης αυτή τη στιγμή διεξάγουν μία έρευνα σχετικά με την οικονομική κατάσταση. Πιστεύω πως θα έπρεπε να συμπεριληφθεί και αυτή η έρευνα στον εσωτερικό κανονισμό. Είναι πολύ σημαντική για να μείνει εκτός. Ε, μετά πιστεύω ότι και η έρευνα για το ΑΕΠ θα μπορούσε να συμπεριληφθεί. Χρειάζεται μία μελέτη που να καλύπτει ευρύτερα θέματα, την κατανάλωση για παράδειγμα, τον ε, πλούτο. Η έρευνα ΣΥΛΚ καλύπτει πολλά από αυτά και θα επέτρεπε μια καλύτερη, ενδελεχέστερη ανάλυση του πλούτου στα νοικοκυριά. Θα συμπεριλαμβάνε, πιστεύω, και άλλους ε, μακροοικονομικούς δείκτες έτσι ώστε να μετρήσουμε καλύτερα το τι γίνεται στα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κανονισμός αυτός ε, τώρα λέγεται ότι θα τεθεί σε ισχύ το 2019. Πιστεύω πως είναι πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα αυτό. Πρέπει να εξετάσουμε τις τροπολογίες που ζητούν παράταση να τεθεί σε ισχύ το 2020-2021, διότι έτσι θα έχουμε αρκετό χρόνο έτσι ώστε να διασφαλίσουμε πραγματικά την θέση ισχύ ενός πλήρως λειτουργικού κανονισμού. Τώρα, για όσους ε, έχουν εκφράσει ανησυχίες γι' αυτό, να, ε, να πω πως ε, τους στηρίζω. Και σε ό,τι αφορά την επικουρικότητα, έχουμε καθήκον να διασφαλίσουμε έναν δυνατό προοδευτικό κανονισμό. Και η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων είναι κάτι που θα βοηθήσει όσους χαράσουν πολιτική διότι αντικατοπτρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Πρέπει λοιπόν αυτές να ποσοτικοποιηθούν έτσι ώστε να ξέρουμε τι συμβαίνει. Ευχαριστούμε πολύ κύριος Ρομπέρο φορ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω Πρώτα απ' όλα μετά από τα όσα μας ανέφερε ως τροπολογής του Συμβουλίου ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, οι στοιχεία που συζητώνται στην ομάδα ε, του Συμβουλίου. Ε, σε σχέση με αυτά λοιπόν, ε, πρέπει να πω ότι δεν εκπλήσωμε που αναρωτιόμαστε για τις προθεσμίες. Είναι μεγάλες αυτές οι προθεσμίες ε, και προσπάθησε να εξισορροπήσει την ευελιξία και τα χρονοδιαγράμματα ε, σαν να χρειαζόταν ε, να αφήσουμε μπόσκα και να έχουμε περισσότερη ευελιξία για να μπορέσουν να τηρηθούν οι προθεσμίες. Και έγινε και μια αναφορά στο Ευρωπαϊκό Εξάμενο. Ναι, πιστεύω και εγώ ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμενο ε, θα πρέπει να αξιοποιήσει οικονομικά και κοινωνικά στατιστικά στοιχεία και κοινωνικά στοιχεία, όχι μόνο οικονομικά, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνει εις βεαρός της ποιότητας, της συγκρισιμότητας, ε, δηλαδή πρέπει να γίνει σοβαρή δουλειά. Η στατιστική που είναι το πρώτο μου επάγγελμα που εξεξά για 30 χρόνια είναι επιστήμη. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η επιστημονική σκέψη που καθορίζει τις προϋποθέσεις από τις οποίες πρέπει να γίνεται η στατιστική ε, θα πρέπει να πέσουν θύμα της ε, ταχύτητας και της ευελιξίας. Ε, στις έρευνες ε, για τους προϋπολογισμούς ε, των οικοκυριών πράγματι ήταν μεγάλα τα χρονικά διαστήματα και για τον εναρμονισμό, για την εναρμόνιση αυτών των ερευνών. Αυτές οι έρευνες, ξέρετε, είναι από τις πλέον πλούσιες που υπάρχουν. Το να ψάξει να βρει κάποιο πώς ζουν, πώς καταναλώνουν, πώς ξοδεύουν χρήματα οι οικογένειες, πώς αποταμιεύουν. Ε, εδώ λοιπόν μιλάμε για μια επιστήμη όπου πρέπει να ακούσουμε τι έχει να μας πει η Συμβουλευτική Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για τις στατιστικές. Ε, ε, ιδρύθηκε πριν από μερικά χρόνια, αρκετά πολλά χρόνια και πρέπει να τους ακούσουμε. Τώρα για τα όσα είπε ο συνάδελφος Ερήκε προηγουμένως, ε, αναφέρθηκε στη στατιστική σαν μια ε, ε, άλλη μορφή του ψέματος. Εγώ θα έλεγα ότι αποτελεί μάλλον αντανάκλαση. Ε, σαν ένας αλκοολικός που ψάχνει τα κλειδιά που έχασε που έχασε κάτω από μια λάμπα στον δρόμο και ψάχνει κάτω από τη λάμπα γιατί εκεί έχει φως χωρίς απαραίτητα τα κλειδιά να έπεσαν κάτω από τη λάμπα. Οι στατιστικές λοιπόν είναι κάπως έτσι. Ε, πρέπει να ξέρουμε πού θα βάλουμε το φως. Τι ακριβώς θα είναι αυτό το οποίο θα εξετάσουμε ε, και κατά πόσο αυτό αντιστοιχεί σε πολιτικές προτεραιότητες. Ε, αλλά τις πολιτικές προτεραιότητες που πραγματικά θέλουμε, όχι αυτές που αναγκαζόμαστε. Η άσκηση αυτή λοιπόν χρειάζεται χρόνο και πολλές προσπάθειες. Συμφωνώ δηλαδή με αυτά που υπόθηκαν για τα νοικοκυριά, αλλά θα ήθελα να μου απαντήσει η Κομισιόν το εξή. Δεδομένων των όσων είπε και η, η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Στατιστικές, ε, υπάρχει, υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία δεν φωτίζουμε αρκετά νωρί ώστε να δούμε μετά από μερικά χρόνια τι γίνεται. Και εκεί τίθεται και το θέμα των νοικοκυριών δεδομένου ότι κοινωνικά μεταβάλλονται σημαντικά. Οι τρόποι ζωής αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε χρειαζόμαστε έναν ορισμό των οικοκυριών που να λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη των διαφόρων μορφών ε, διαβίωσης. Μετά έχουμε το ζήτημα της μετανάστευσης επίσης και το πολύ μικρό άνοιγμα στα θέματα του περιβάλλοντος. Δηλαδή στο πώς έχουμε διάφορους τρόπους ε, διαβίωσης ε, ε, περιβαλλοντικούς για να πούμε έτσι. και επίσης ε, έχουμε τις απογραφές που ρυθμίζονται από άλλο κανονισμό. Ε, ούτε αυτές πρέπει να τις ξεχνάμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πέντε λεπτά. γνωρίζοντα ότι σα έγιναν πολλές ερωτήσεις, ε, φαντάζομαι θα μπορέσετε σε πέντε λεπτά κάπως να μα ε, διαφωτίσετε κάπω. Thank you, uh, thank you, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τα πολύ χρήσιμα σχόλια και για τη στήριξή σας, αλλά και τις ερωτήσεις. Λοιπόν, μερικά στοιχεία τώρα. Κατά πόσο ο κανονισμός αυτός είναι συμβατός ε, με το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα και άλλα κείμενα. Ναι, αλλά οπωσδήποτε πρέπει όλα αυτά να είναι συμβατά. Ό,τι κάνουμε πρέπει να εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο. Και να μην ε, συγκρούεται με άλλους κανονισμούς. Το σημειώνω. Είναι απόλυτα σαφές. Πρέπει έτσι να είναι. Τώρα, Υπάρχουν ε, μια σειρά από ορισμοί που έχουν προταθεί. Φυσικά ο στόχος του άρθρου 2 του κανονισμού δεν είναι να κάνει ένα μακρύ κατάλογο στατιστικών όρων, να διατυπώσει ένα μακρύ κατάλογο στατιστικών όρων. Θέλουμε μόνο τα πιο ουσιώδη, τα πιο ουσιώδη για να διασφαλίσουμε την πιο σωστή εφαρμογή του κανονισμού. Ορισμένοι από τους, ορισμοί που προτείνονται, από τους ορισμούς που προτείνονται είναι πολύ καλοί. Κάποιους άλλους πρέπει να τους ξαναδούμε. Και πρέπει να περιοριστούμε μόνο στους απολύτως ε, αναγκαίους ορισμούς. Ορισμένοι θα μπορούσαν, εάν προσθεθούν όμως, να δημιουργήσουν ε, μία μείωση της αφήνειας. Βεβαίως και πρέπει επίσης να συμμορφούμεθα με τον κώδικα στατιστικής διοντολογίας. Βεβαίως και αυτό το σημειώνω και είναι προφανές. Τώρα κατά πόσο είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος αυτός ο κανονισμός και ιδιαίτερα πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται, προβλέπουμε το 19. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου εργαζόμεθα σε αυτή τη φάση. Αλλά σημειώνουμε τι είπατε. Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος και η κοινή τους κατανομή. Ναι, τα στοιχεία πλούτου θα είναι στον κανονισμό. Όχι όλος ο πλούτος, όλα τα περιουσιακά στοιχεία γιατί συνεργαζόμεθα πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που επίσης ε, ε, ε έχει αυτή την έρευνα για τα περισσοκά στοιχεία σε συνεργασία με τις, Ευρωπαϊκές, με τις ε, Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Φυσικά δεν θέλουμε επικάλυψη προσπαθειών με την ΕΚΤΑΦ. Διεθνή συγκρισιμότητα. Και αυτό είναι πολύ βασικό στοιχείο. Οι ορισμοί μας, ε, οι αντιλήψεις μας είναι ταυτόσιμοι με τους αντίστοιχους ορισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Άρα είναι διασφαλισμένη η διεθνή συμβατότητα. Τώρα βέβαια λέμε ότι η ταχύτητα συλλογής των στοιχείων, η ποιότητα και η συγκρισιμότητα όλα αυτά μπορεί να αντιβαίνουν λιγάκι το ένα το άλλο. Προσπαθούμε να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία, ούτω ώστε τα στοιχεία μα και να έχουν έννοια και να μην καθυστερούν πολύ σε σχέση με τι ανάγκε. Πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν για να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία. Τώρα το, την έρευνα για το προπολογισμό των οικοκυριών βεβαίω είναι μεγάλη σημασία. Χρησιμοποιείται και για του εθνικού λογαριασμού, για τι τιμέ, για το καλά τιμών. Βεβαίω είναι πολύ σημαντική αυτή η έρευνα. Αλλά από τώρα μέχρι το τέλος της δεκαετής ε, περίοδου αυτές οι έρευνες για τον προϋπολισμό των οικοκυριών θα συνεχίσουν να γίνονται από τα κράτη, δεν θα τις σταματήσουμε. Απλώς τις εξυγχρονίζουμε. Θέλω επίσης να σας ε, διαβεβαιώσω ότι λαμβάνουμε υπόψη την κοινωνική διάσταση. Ε, νέοι τρόποι ζωής, νέα φαινόμενα, μετανάστευση, ένταξη, περιβάλλον ιδιαίτερα. Δηλαδή συνθήκες και ποιότητα ζωής. Τα λαμβάνουμε υπόψη. Και συνοηθήκαμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΖΑΚ όπως τη λέμε, και λάβουμε υπόψη την ε, γνωμοδότηση που μας έδωσαν. έγινε η παρατήρηση ότι το στατιστικό στοιχείο αγορά, ε, συγγνώμη, εργατικό δυναμικό θα πρέπει να αντικατασταθεί από την αγορά εργασίας. Ε, εργατικό δυναμικό είναι οι εργαζόμενοι συν άνεργοι, αλλά καλύπτουμε και άλλους τους ανενεργούς κτλ. Θέλουμε να έχουμε μια ευρύτερη έννοια εδώ για το τι σημαίνει αγορά εργασίας. Γι' αυτό Γι' αυτό το αποκαλούμε εργατικό δυναμικό, ενώ στην ουσία είναι αγορά εργασία. Και καλύπτουμε βεβαίω έτσι και την ε, δραστηριότητα των επιχειρήσεων μέσω ακριβώ τη έρευνά μα για τι επιχειρήσει. ΝΑΤΣ 2, περιφερειακά και πιο τοπικά στοιχεία, βεβαίω είναι πολύ σημαντικό. Είναι δύσκολο τομέα γιατί μπορεί να έχει μεγάλο κόστο. Βεβαίω, συμφωνούμε ότι πρέπει να δίνεται στο σωστό επίπεδο η προφορία αλλά πρέπει να είναι και συγκρίσματα στοιχεία. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια μελέτη εφικτού και μετά από αυτές τις μελέτες θα επιχειρήσουμε να έχουμε τα στοιχεία σε επίπεδο NATS 2. Αυτά νομίζω σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις αυτές. Λοιπόν, προθεσμία υιοθέτηση στην Επιτροπή 29 και 30 Μαΐου. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Έλεγχο δαπανών και παρακολούθηση της οικονομικής αποδοτικότητας των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωση ε, Εγγύηση για την Νεολαία. Σας δίνω αμέσω το λόγο ε, δεν είναι εδώ η συγκήτρια, οπότε δίνω το λόγο στην κυρία Τρεμπίσους για τέσσερα λεπτά, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρους της ε, συναδέλφου Γιάννα Τινάνσκα, η συγκήτρια του ΙΣΙΑΡΑ. Η Επιτροπή μας φέτος θα αφιερώσει τεράστιες προσπάθειες σε προγράμματα με στόχο τους νέους για τις δεξιότητές τους και την απασχολησιμότητά τους. Αναμένουμε μια πλήρη έκθεση υλοποίησης που ονομάζεται η υλοποίηση της ε, πρωτοβουλίας ε, εγγύηση για την νεολαία στα κράτη-μέλη. Ε, η γνωμοδότησή μου για την εγγύηση για την νεολαία και την παρακολούθησή της ε, αναφέρει ότι πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της εγγύσης για την νεολαία και της ε, πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Ε, εγώ θα προσπαθήσω να τηρήσω την εντολή αυτής της γνωμοδότησης, να σας πω τι θεωρώ σημαντικό και τι προσπάθησα να εντάξω στο σχέδιο του κειμένου. Πρώτα απ' όλα, η εγγύηση για την νεολαία θεωρώ ότι είναι μια πολιτική δέσμευση και σοβαρή προσπάθεια μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Με ένα σύνολο εγγυήσεων για το νεολαία, τα κράτη-μέλη συμφωνούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους νέους, ώστε οι ικανότητές τους να μην σπαταλώνται. Η εγγύηση για την νεολαία σήμερα εξαρτάται από τις προϋπάρχουσες δυνατότητες που υπάρχουν στα κράτη-μέλη στις υπηρεσίες απασχόλησής τους για να φέρουν αποτελέσματα για τους νέους. Γι' αυτό το λόγο ενθαρρύνω τα κρατημέλη να κάνουν περισσότερα για να υλοποιήσουν ε, την εγγύηση για την νεολαία μέσω ε, δημιουργίας εταιρικών σχέσεων, συνεργασιών, ε, βελτιώνοντας οι και, μέσω, και δημιουργώντας τις σωστές δομές αξιολόγησης. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι για να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό του σχεδίου αυτού δεν πρέπει να ξεχνάμε τις πιο ευάλωτες ομάδες ε, διαφοροποιημένες, μεμονωμένες προσεγγίσεις όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών στους νέους ανθρώπους που τις χρειάζονται περισσότερο ώστε να αποφεύγονται οι ε, ε, διαλογές έτσι όπως ονομάζονται. Πολλοί από εσάς έχουν δει τα αποτελέσματα της τελευταίας έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου που δημοσιεύτηκε την, την περασμένη εβδομάδα. εγώ θα συμπεριλάβω και στοιχεία που αφορούν τα αποτελέσματα της εγγύησης για τους νέους ε, και θα αναμένω τις προτάσεις σας για να συνεχιστούν οι συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για το έλκη Σοφία Ριμπέρο ε, στη θέση της κυρίας Ενιάς Κακόλοφσκα για το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ. Θα διαβάσω τη δήλωση της κυρίας Κοσλόσκα οι επιδόσεις των νέων στην αγορά εργασίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά από το 2013. 14 εκατομμύρια νέοι είχαν πρόσβαση στην εγγύηση για τους νέους και 9 εκατομμύρια δέχτηκαν προσφορά εργασίας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η εγγύηση για τους νέους έχει γίνει κινητήριος δύναμη για το εργατικό δυναμικό και ε, βοήθησε στην αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της εκπαίδευσης. Τα προγράμματα ωστόσο του, της για τους νέους δεν έχουν φτάσει σε όλους τους νέους ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει πολλές φορές το σχολείο. Υπάρχουν λοιπόν ε, ορισμένοι τομείς που επιδέχονται βελτίωσης. Καταρχάς η απασχολησιμότητα πρέπει να ενισχυθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί ομαλή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη ακόμα δεν έχουν κάνει εντελεχείς αναλύσεις που θα τους επιτρέψουν να δουν ε, τις ανάγκες του πληθυσμού. Υπάρχουν πολλές φορές ε, λάθος εκτιμήσεις και γι' αυτό η εγγύηση για τους ε, νέους μπορεί να βοηθήσει. Δύο, εντοπισμός ε, αναγκών που δεν έχουν καταγραφεί. Τα κράτη-μέλη έχουν ανάγκη εντοπισμού αυτών των αναγκών. Γι' αυτό η σκέδα συγγήτρια θα ήθελε να εστιάσει στις ανάγκες που δεν έχουν καταγραφεί και δεν καλύπτονται από το εφιστάμενο σύστημα για ορισμένες ομάδες. Ε, καλή για στενότερη συνεργασία των ενδιαφερόμενων φορέων, δημόσιου ιδιωτικού τομέα, υπηρεσιών έβρεσης εργασίας, ε, ιδρυμάτων ε, εκπαίδευση κατάρτισης. Τρίτον, μείωση διοικητικού άχθους γραφειοκρατία είναι υψηλή, γι' αυτό χρειάζεται να ληφθούν μέτρα τα οποία θα διασφαλίσουν πως οι νέοι θα λαμβάνουν μία προσφορά εργασίας ε, ποιοτική, ε, μία ποιοτική επίσης ε, θέση μαθητείας, έτσι ώστε να αποφύγουν το να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο και να μείνουν άνεργοι. Μετά, ο Σκιώδης συζητητή έχει ένα σχόλιο για την παράγραφο 6 της νομοδότησης, η οποία εφιστά την προσοχή ε, απέναντι ε, στους κινδύνους μη διάδοσης ε, του προγράμματος εγγύηση για τους νέους. Χρειάζεται οι νέοι να λαμβάνουν ποιοτικέ προσφορές οι οποίες να είναι προσαρμοσμένες στις δικές τους δεξιότητες και ανάγκες. Αυτό βέβαια θα υποβληθεί και ως τροπολογία. Η κυρία Κοσλόφσκα θα χαρεί πολύ για τη μελλοντική συνεργασία με την εισηγήτα και όλους και όλες εισηγητές και ε, σας ευχαριστώ ξανά για την γνωμοδότηση. Ευχαριστούμε πολύ για το η κυρία Μαρτίνα Δαγιολοβά. Ε, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συναδελφοί. Πρέπει να πω ότι η συναδελφός έγραψε μια εξαιρετική γνωμοδότηση και θέλω να την ευχαριστήσω. Και εγώ είχα το προνόμιο να εργαστώ στο ίδιο ζήτημα τόσο από την άψη τη δημοσιονομική όσο και από την άψη τη απασχόληση. Τώρα έρχομαι από την εποχή έλεγχου του προπολογισμού όπου συζητήσαμε μια νέα ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου που αναφέρθηκε ήδη και που ονομάζεται απασχόληση των νέων κατά πόσο οι ευρωπαϊκές πολιτικές έκαναν μια διαφορά και τι γίνεται με τις δύο πρωτοβουλίες ε, απασχόλησης και εγγύησης για την νεολαία. Οπότε είναι καλό που θα έχουμε την ευκαιρία στις 25 Απριλίου να συζητήσουμε με την κυρία Ιβάνοβα για την ειδική έκθεση. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι μερικές φορές βλέπουμε τα πράγματα από διαφορετικές ε, ε, οπτικές γωνίες στην Επιτροπή Απασχόλησης και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να εντάξουμε και τις δύο αυτές οπτικές γωνίες όλες τις εκθέσεις που θα γράψουμε. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ε, τα κύρια ευρήματα, τι βλέπουμε εμείς από την ε, άψη του ελέγχου του προπολογισμού ως ε, σημαντικό. Πρώτον, το ελεγκτικό συνεδρίο στην έκθεση αυτή έκανε μια πολύ καλή στατιστική έρευνα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και τι πληροφορίε που συλλεγήσαν και σε αυτή την εδώ την έκθεση. Ε, όχι μόνο δεν βρήκαμε λάθη στις δαπάνες των ταμείων αυτών, όχι μόνο συγγνώμη, θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τα λάθη, αλλά θα πρέπει να δούμε και πώ μπορούμε να τα αποφύγουμε στο μέλλον. Γιατί με αυτά τα πολύπλοκα προγράμματα πολλέ φορέ τα ίδια λάθη επαναλαμβάνονται διαρκώ. Οπότε πρέπει να μαθαίνουμε από το παρελθόν. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό και χαίρομαι που το έχουμε συμπεριλάβει στην γνωμοδότησή μα. Θα πρέπει να αναπτύξουμε ε, βέλτιστες πρακτικές και να τις συζητάμε γιατί ξέρετε πολλές φορές μιλάμε, λέμε βέλτιστες πρακτικές αλλά δεν τις ε, ε, χρησιμοποιούμε πραγματικά δεν τις αξιοποιούμε κάποιες βελτιστές πρακτικές που έχουν επιτυχία σε κάποιες περιφέρειες, σε κάποια κράτη-μέλη, χωρίς να έχουν διαδοθεί σε άλλες χώρες. Οπότε αυτό πρέπει να το προωθήσουμε. Κάτι άλλο σημαντικό είναι να ορίσουμε ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους, καθώς και μετρήσιμους στόχους. Ε, αυτό είναι ενδιαφέρον. Ε, το ανέφεραν κάτι συνάδελφοι. Έγινε μια συζήτηση στην Επιτροπή Ελεκτού Προπολογισμού, μάλιστα, για το τι σημαίνει καλή ποιότητα προσφοράς, ε, μια προσφορά καλής ποιότητας. Από ευρωπαϊκή άποψη η προσφορά αυτή καλής ποιότητας τι σημαίνει, σημαίνει προσφόρα εργασίας που ταιριάζει με τις ικανότητες του συμμετεχόντος και που βοηθά στο να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Μ' αρέσει αυτός ο ορισμός γιατί μας έλειπε ένας ορισμός και είμαι πεπισμένη ότι μια καλή προσφορά είναι κάτι πολύ ατομικό, εξαρτάται από το συγκεκριμένο πρόσωπο, ποτέ πρέπει να προσέξουμε πώς θα το μετρήσουμε. Τελευταίο που ήθελα να αναφέρω και θεωρώ ότι είναι σημαντικό, που πιστεύω ότι πρέπει να προωθήσουμε και από την Επιτροπή Απασχόλησης, είναι η συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, διότι μερικές φορές τα προβλήματα υλοποίησης της ε, ε, εγγύησης για την νεολαία εμφανίστηκαν λόγω κάποια συμφωνία μεταξύ ε, εθνικού, περιφερειακού και ευρωπαϊκού επίπεδου. Χρειάζεται λοιπόν τεχνική ε, αρρωγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κρατημέλη και τις περιφέρειες. Αυτή είναι η κατεύθυνση ε, προς την οποία θα κινηθούν οι τροπολογίες που θα υποβάλω για να υπογραμμίσω αυτές τις συστάσεις. Αλλά είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με τη δουλειά της Γιάννα Ζητνιάνσκα Μ' αρέσει που βλέπουμε το θέμα αυτό με τόσο ολιστικό τρόπο στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την ΚΟΕ, η κυρία Λοπές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεύτερη φορά που το ελεγκτικό συνέδριο ε, μας τη λέει. Πρώτα για το ΕΦΣΙ και τώρα με την εγγύηση για τους νέους. Γιατί δεν λειτουργεί σωστά το πρόγραμμα, είναι προφανές. Σίγουρα είναι αναγκαίο, δεν το αμφισβητώ. Γιατί λόγω της λιτότητας που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ευρωπαϊκά ταμεία είναι μία από τις λίγες πηγές που επιτρέπουν τη χρηματοδότηση για την απασχόληση. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, τα ταμεία αυτά εφίστανται αλλεπάλληλες περικοπές στους προπολογισμούς τους. Και επιπλέον, δεν υπάρχει κανένα έλεγχος για την ε, ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρεται, ούτε για τον προσανατολισμό, ούτε για το είδο ε, εκπαίδευση, ούτε τα συνοδευτικά μέτρα, ούτε για το εάν περιλαμβάνονται οι πιο ευάλωτε ομάδε. Και σίγουρα ένα τμήμα αυτών των ε, χρηματοδοτήσεων στην ουσία είναι επιδότηση για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τους νέους ως φτηνή εργατική δύναμη που τη χρησιμοποιούν όσο λαμβάνουν επιδότηση και μετά την ε, απολύουν. Πρέπει φυσικά να αλλάξει τρόπος, ε, ο τρόπος χρήσης. Πρέπει να συμμετέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες, πρέπει να συμμετέχουν τα συνδικάτα. Έτσι μόνο θα αναπτυχθεί αυτή η πρωτοβουλία στα κράτη-μέλη και στις αυτόνομες περιφέρειες ή τις περιφέρειες των κάποιων κρατών. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τους νέους εργαζόμενους. Και δεν θα σταματήσω να λέω. Το πρόβλημα της ε, ανεργίας των νέων είναι πάνω απ' όλα διαρθρωτικής φύσης, μακροοικονομικό. Οπότε, εκτός από αυτό το πρόγραμμα, πρέπει επίσης να υπάρξουν περισσότερες δημόσιες επενδύσεις, να αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής και να ενισχύσουμε και τη δυνατότητα συλλογής φόρων για να υπάρξουν αναδιανεμητικές πολιτικές. Μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά η εγγύηση για τους νέους και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των νέων μας που δυστυχώς υποφέρουν τις χειρότερες επιπτώσεις της χειρότερης περίοδου ανεργίας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και η κυρία Τέρι Ρένκεν για τους πρασίνους. Ευχαριστώ και εγώ την ε, εισηγήτρια. Ανέφερε πολλά σημαντικά σημεία που πρέπει και εμείς να τα τονίσουμε στη συζήτηση για την ε, παρακολούθηση του προγράμματος για την εγγύησεων για την νεότητα. Κάτι που κατέστη απόλυτα σαφές και στην ακρόαση που κάναμε πριν από τρεις ε, εβδομάδες εδώ και μετά και την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε, επειδή είμαστε στις αρχές ακόμη, δεν μπορούμε να προτρέξουμε τώρα, να εξαγάγουμε δεν έχουμε ακόμη τις στατιστικές. Όμως πρέπει να το παρακολουθούμε στενά. Πρέπει να ελέγξουμε πώς δαπανούμε τους πόρους αυτούς, αλλά και για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το πρόγραμμα αυτό εγγύησεων για την νεότητα για να επιτύχει ουσιοδός. Συμφωνώ με ορισμένου συναδέλφου που είπαν ότι είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση εφαρμογή από κράτο μέλο σε κράτο μέλο. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και σε όποια κράτη-μέλη δεν τα πάνε καλά, πρέπει να τονίσουμε ότι θέλουμε βελτίωση. Τώρα, όπως είπε και η κυρία Ζιντάνσκα στο σημείο 4, και εγώ θέλω να τονίσω ότι πρέπει να είναι πιο στοχευμένα προς συγκεκριμένες ομάδες νέων αυτά τα μέτρα, γιατί πολύ συχνά τι βλέπουμε, Οι προτάσεις που υποβάλλονται απευθύνονται μόνο σε ορισμένες ομάδες νέων που είναι αυτοί στους οποίους μπορούμε να απευθυνθούμε πιο εύκολα. Το βασικό είναι όμως να έχει αντίκτυπο και στις πιο ευάλωτες ομάδες νέων αυτό το πρόγραμμα. Και κάτι άλλο που θα υποβάλουμε και μέσω τροπολογιών, η εγγύηση για την ενότητα θα πρέπει να καταπολεμήσει την ε, ανεργία των νέων αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας των κρατών μελών. Αυτό πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Από μόνο του το πρόγραμμα αυτό, μαζί με την πρωτοβουλία για την ε, απασχόληση των νέων, δεν μπορεί να διορθώσει τα λάθη που έχουν διαπραχθεί στην ε, μακροοικονομική πολιτική. Όταν επικρίνουμε τον τρόπο εφαρμογή του στα κράτη-μέλη, θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να αλλάξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για τι μακροοικονομικέ πολιτικέ, ούτω ώστε το πρόγραμμα αυτό να επιτύχει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Λοιπόν, προθεσμία για τις τροπολογίες, 25 Απριλίου, 12 το μεσημέρι. Θα το εγκρίνουμε είτε στις 22 είτε στις 21 στις 22 Ιουνίου και θα εγκριθεί από την Αρμόδια Επιτροπή 12-13 Ιουλίου και κατά πάσα πιθανότητα αργότερα από την Ολομέλεια. Θα τα ξαναπούμε στις 25 Απριλίου. Νομίζω ότι είναι η εθνική ορδή τη Πορτογαλίας, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ε, σας εύχομαι να περάσετε καλά. Καλή Ανάσταση.